Good morning, colleagues. Um, we begin this morning with... Καλημέρα, συνάδελφοι. Ξεκινάμε αυτή τη συνεδρίαση. Μετά από τι τρομοκρατικέ επιθέσει στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου, υπό την παρουσία τη Προεδρία ε, του Συμβουλίου, στην τελευταία μα συνεδρίαση συζητήσαμε το θέμα αυτό των ε, Βάρβαρ βάρβαρων επιθέσεων στο Παρίσι και σήμερα θα έχουμε λοιπόν και μια ενημέρωση από την ε, Λουξεμβουργιανή Προεδρία για τη θέμα αυτό και σε σχέση με τα αποτελέσματα της, ε, του σχετικού συμβουλίου της, ε, του Συμβούλου GAG. Μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Κίρκοπ να μας ενημερώσει για το σημαντικό έργο που γίνεται μετά τι επιθέσει, θα γίνει συζήτηση και ανάλυση αυτών και τέλος θα δώσω τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα γίνουν ανταλλαγέ απόψεων με την Europol, με την Interpol στι επόμενες συναντήσεις μας. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στο κύριο Λιμπρέκεν από την Λουξεμβουργιανή Προεδρία. Έχετε το λόγο. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που δίνετε στην Προεδρία την ευκαιρία να σας παρουσιάσει εν συντονία, συντομία τα πρεπραγμένα του Συμβουλίου Τζάι που έλεγε χώρα τον ε, Νοέμβριο. Πριν να περάσω σε λεπτομέρειες όσον αφορά τις εργασίες του Συμβουλίου, επιτρέψτε μου καταρχάς να υπογραμμίσω το συμβολικό χαρακτήρα που είχε η διεξαγωγή αυτού του Συμβουλίου μία εβδομάδα μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι. Το Συμβούλιο αυτά, αυτό χρησιμεύσε καταρχάς για να δείξει την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τη Γαλλία και να δείξει και την ενότητα της Ένωσης ενώπιον τέτοιων αποτρόπεων πράξεων. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το Συμβούλιο όχι μόνο συγκέντρωσε τους Υπουργούς Εσωτερικών αλλά και τους Υπουργούς Δικαιοσύνης. Πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα σημαντικό μήνυμα για να δείξουμε ότι ο τομέας των εσωτερικών και ο τομέας της δικαιοσύνης συνεργάζονται στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το Συμβούλιο ενέκρινε, δύο συμπεράσματα. Η πρώτη σειρά συμπερασμάτων αφορούσε την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αυτή καθ' αυτή. Αυτά τα συμπεράσματα συμπεριλαμβάνονται σε μία σειρά από μέτρα, μερικά από αυτά είναι ήδη γνωστά, αλλά τονίζεται πρωτίστως <clears throat> η ανάγκη που υπάρχει να ληφθούν ορισμένα μέτρα και δράσεις από πλευράς της Ένωσης. Το πρώτο στοιχείο επί του οποίου οι Υπουργοί επέμειναν αφορούσε την όσο το δυνατόν ταχύτερη έγκριση της οδηγίας για το, σύστημα, για το Ευρωπαϊκό Σύστημα PNR. Κατά τη διάρκεια του γεύματος οι Υπουργοί μπόρεσαν να συνομιλήσουν με τον Πρόεδρό σας σχετικά με το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Το άλλο θέμα που συζητήθηκε και που συμπεριλήφθη στα συμπεράσματα αφορούσε τα όπλα, ο έλεγχος των όπλων. Δηλαδή, οι υπουργοί χαιρέτησαν την έγκριση ενός κανονισμού για τους κοινού κανόνες σε ό,τι αφορά την εξουδετέρωσή τους και θα πρέπει να χαιρετήσουμε το γεγονός ότι η Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση που στόχο είχε την αναθεώρηση των όπλων. Νομίζω ότι και η Επιτροπή θα, πει για λόγια για αυτό το θέμα μετά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα, οι Υπουργοί ανέλαβαν τη δέσμευση να εξυγχρονίσουν μέχρι το Μάρτιο του 2016 το σύστημα ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση με τη βάση σχετικών δεδομένων, ιδιαίτερα με τα δεδομένα της Ιντερπόλ. Στα πλαίσια της ε, μεταναστευτικής κρίσης ελήφθη η δέσμευση να διεξάγεται συστηματικός έλεγχος ασφαλείας των ρευμάτων που εισέρχονται στην κοινότητα ελέγχοντας τα, τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένα, δεδομένων της Ένωσης και της Ιντερπόλο. Οι υπουργοί, στα πλαίσια του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων, τόνισαν και πάλι το γεγονός ότι θεωρούν ότι είναι αναγκαίο όπου υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν ε, ομάδες ε, άμεσης επέμβασης της Frontex. Οι Υπουργοί έκαναν έκκληση στην Επιτροπή να επανεξετάσουν τον κώδικα των συνόρων Σέγγεν με στοχοθετημένο τρόπο έτσι ώστε να ελέγχεται ε, να ελέγχονται τα σύνορα. Υπήρξε επίση μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Υπουργών και μια ανάληψη δέσμευσης έτσι ώστε η εθνικές αρχές το SES2 να συμπεριλάβουν στοιχεία που αφορούν τους ξένους μαχητές, του υποτιθέμενους ξένους μαχητές για να μπορέσουν να, ε, για να μπορούν να εντοπίζονται το συντομότερο δυνατόν όταν μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Υπουργοί ανέλαβαν τη δέσμευση να εφαρμόσουν άμεσα και στο σύνολό του το κεκτημένο. Χαιρέτησαν το γεγονός ότι η Europol θα ήδη στο κέντρο καταπολέμησης της δημοκρατίας. Πιστεύω ότι ο διευθυντής της Europol, ο κύριος Winwright, είχε την ευκαιρία να σας μιλήσει για αυτό το θέμα την προηγούμενη εβδομάδα. Θα επιθυμούσα κυρίως στα πλαίσια της ανταλλαγής αυτής πληροφοριών να υπογραμμίσω ότι πραγματικά Όλοι συμφώνησαν ότι θα πρέπει να ενδυναμωθούν τα υπάρχοντα μέσα και η Προεδρία ανέλαβε την υποχρέωση να επανέλθει στο θέμα αυτό και την Παρασκευή θα διεξαχθεί μια λεπτομερής συζήτηση μεταξύ των Υπουργών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διαφόρων στοιχείων του κεκτημένου που υπάρχει σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών. Το Συμβούλιο ασχολήθηκε με το, θέμα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υπογραμμίζοντας το ρόλο που παίζουν ε, οι ε, πυρήνες, οι ομάδες χρηματοδότησης και είπαν ότι στόχος ήταν να εναρμονιστεί ο συντονισμός αυτών των μονάδων οικονομικών πληροφοριών. Οι υπουργοί κάλεσαν την Επιτροπή και ελπίζω να ανταποκριθεί άμεσα να υποβάλει μια αναθεώρηση του ποινικού πλαισίου της ε, απόφασης πλαισίου που αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας για να μεταγραφεί στην Ένωση το ε, συμπληρωματικό πρωτόκολλο της σύμβασης που αφορά την πρόληψη της τρομοκρατίας, σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μετά οι Υπουργοί κάλεσαν την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες της σε ό,τι αφορά το σύστημα ε, ε, πληροφοριών σχετικά με το ποινικό μικρό. Κατόπιν οι Υπουργοί οθέτησαν με άλλη σειρά από συμπεράσματα σχετικά με το θέμα της ριζοστικοποίησης, ριζοσπαστικοποίησης. Η Επιτροπή στο σύνολό της με την Προεδρία οργάνωσαν μία εκτενή συζήτηση για το θέμα αυτό τον Οκτώβριο. Τα συμπεράσματα αυτά αποτελούν καρπό αυτής της εργασίας. Λαμβάνονται υπόψη τα όσα έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η και πιστεύω ότι είναι σημαντικό σε αυτόν τον τομέα να κινηθούμε από κοινού Μολονότι είμαστε σε ένα τομέα όπου κατά βάση οι χώρες μέλη είναι εκείνες ε, που χειρίζονται την κατάσταση γιατί είναι εκείνες υπεύθυνε για την διαχείριση των φυλακών. Είναι δηλαδή θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των χωρών μελών. Αυτό βεβαίως δεν εμποδίζει να γίνει κάτι σημαντικό σε επίπεδο ένωσης, σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική δουλειά για να υπογραμμίσουμε το ρόλο που παίζει η πρόληψη μιλώντας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, με λίγα λόγια, αυτά συζητήθηκαν από τους υπουργού Εσωτερικών και Δικαιοσύνης την προηγούμενη εβδομάδα σε συνέχεια των επιθέσεων στο Παρίσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα περνάμε στον κύριο Κέρκοφα ε, κατευθείαν από την ε, Επιτροπή Αντιτουρομοκρατικών Μέτρων μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο καθότι η Πρόεδρια υπήρξε σε μεγάλο επίπεδο λεπτομέρειας σε σχέση με τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει από τις επιθέσεις του Παρισιού και μετά να αναλύσω κάποιε συγκεκριμένε ψυχέ. Καταρχά τα πρόσφατα περιστατικά, όχι μόνο στο Παρίσι, αλλά και στην ε, Άγκυρα, πάνω από 100 νεκροί, στο Σινάι, 230-240 στην ε, σε Τιμίδα και Παρίσι. Όλα αυτά υποδεικνύουν ε, την δραστηριότητα της του Ισλαμικού κράτους που ως τώρα προσπαθεί να δημιουργήσει το χαλιφάτο και έχει βάλει στο στόχαστρο τα μέλη της συμμαχίας. Ε, το Ισλαμικό λοιπόν κράτος πάντα προσπαθούσε να δείξει ότι είναι νικητρία, νικητής για να προσελκύσει νέους ε, μαχητές. Και τώρα λοιπόν υπάρχει αντίκτυπο. Και αυτό αναγκάζει ενδεχομένω το Ισλαμικό κράτο να ζητήσει επιτυχίε στο εξωτερικό. Και εδώ λοιπόν αντιμετωπίσουμε τρει προκλήσει, θεωρώ. Καταρχά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταδείξουν στου ε, πολίτε ότι μπορούμε να του προστατεύσουμε. Δεύτερη δυσκολία για την Ευρώπη ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διατηρήσουμε ένα από τα καλύτερα επιτεύγματα της ε, ευρωπαϊκής διαδικασίας ενοποίησης, την ελεύθερη μετακίνηση, το Σέγγεν. Και τρίτον, στο ίδιο πνεύμα, ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ μετανάστευσης και τρομοκρατίας. Είναι τοξικός αυτός ο σύνδεσμος και αυτό προαπαιτεί από όλους μας αποφασιστικότητα ρεαλιστικότητα, πραγματισμό και δράσεις. Όχι πλέον έγγραφα, αλλά δράση. Επιτόπου. Και αυτό λοιπόν προσπαθούν να πετύχουν η Προεδρία του Συμβουλίου τους τελευταίους μήνες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θυμάστε το πλαίσιο, το σημείο αναφορά σε μια δήλωση 12 Φεβρουαρίου των αρχηγών κρατών μετά τις επιθέσεις στην Σαρλή Εμπντο στο Παρίσι και στα καταστήματα που ζήτησε από όλους μας να κινηθούμε προς τρεις κατευθύνσεις. Καταρχάς, κλασική αντίδραση αντιμετώπισης, η οποία και πολύ καλά περιγράφτηκε από τον συνάδελφό μου, αλλά θα τονίσω και κάποιες πτυχές. Κατά δεύτερον, η ήπια αντιμετώπιση, η πρόληψη και η εξωτερική δράση. Για να συμμετέχουν και οι γειτονικέ χώρε, τα Δυτικά Βαλκάνια, η Τουρκία. Θα ήθελα να αντιδράξω λοιπόν αυτέ τι τρει λύσει εν συντομία. Καταρχά, ε, η αντίδραση καταστολή. Να σα πω με ειλικρίνεια η αίσθηση που επικρατεί, και αυτό αναφέρεται και στην έκθεση, και η άποψή μου που μοιράζομαι με την Επιτροπή σα, είναι ότι τα μέτρα τα οποία λήφθησαν το Φεβρουάριο θα έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί πιο γρήγορα και πιο στεναρά. Πολλά είχαν ήδη αποφασιστεί. και ουσιαστικά δύο πτυχές είναι σχετικές. Γεμίζουν τα κάτι μελη τη βάση δεδομένων που έχουμε και την χρησιμοποιούν στο έπακρο. Και το δεύτερο θέμα είναι κατά πόσον είμαστε αρκετά αποτελεσματικοί στα εξωτερικά σύνορα. Κοιτώντα τι έγινε στο Παρίσι, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η απάντηση δεν είναι 100% καταφατική. Ω εκ τούτου, στο Συμβούλιο την ε, προηγούμενη Παρασκευή και την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε αντιμέτωπη με την αλήθεια. Θα εκτιμήσουμε κατά πόσον τα κράτη-μέλη όντως συμπληρώνουν τη βάση δεδομένων, ε, έχουν τα ηλεκτρονικά μέσα, έχουν τις σχετικές συσκευές ανάγνωσης για να το κάνουν αυτό και πιο επίκαιρη βάση δεδομένων, που είναι και το καλύτερο αστυνομικό εργαλείο, είναι το σύστημα ενημέρωσης Schengen, το SIS. Και μέρος των προσπαθειών των τελευταίων μηνών είναι να πείσουμε τις μυστικέ και αστυνομικέ υπηρεσίες να βάζουν στο ΣΥΣ όλα τα στοιχεία που έχουν για τους αλλοδαπούς μαχητές. Είμαστε στην, σε καλό δρόμο και πολλά κράτη-μέλη έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια για την τροφοδότηση του ΣΥΣ με αυτά που ονομάζονται στοιχεία άρθρου 36.3 για τέτοιες ε, μυστικές ε, πληροφορίες. Ε, στη συνέχεια έχουμε και θέματα Interpol. Όταν υπάρχουν στα εξωτερικά σύνορα εξωτερική έλεγχη, ελέγχεται κατά πόσον το διαβατήριο είναι τμήμα της βάσης δεδομένων της Interpol για τα κλαμμένα διαβατήρια, η καλύτερη σχετική βάση σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά η τροφοδότηση θα πρέπει να είναι συστηματική. Και φυσικά, τελευταίο και τρίτο στοιχείο είναι να πείσουμε όλους τους φορείς να συμμετέχουν και να χρησιμοποιούν την Europol, το ECDC, η καλύτερη πλατφόρμα που υπάρχει για το μέλλον, που μπορεί να χρησιμοποιήσει και διάφορα εργαλεία. Το σχένα το οποίο θα αναβαθμιστεί σε δίκτυο εμπιστευτικό το σύστημα πληροφοριών ε, Europol, τα σημεία εστίασης της Europol και όχι μόνο για τέτοια θέματα αλλά και για το trafficking. Το TFTP το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εργαλείο και υποθέτω ότι στην περίπτωση του Παρίσιου το TFTP είχε παρέχει πολλές πληροφορίες ε, στους αστυνομικούς. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία όπως το Internet Refer Unit, τα στοιχεία της Europol, τα συστήματα της Europol για το trafficking και θέλουμε να φτιάξουμε και ένα κέντρο αριστείας. Και είμαι αισιόδοξο ότι αυτά θα χρησιμοποιούνται όλο και πιο πολύ από τα κρατημέλη. Ίσως δύο πρόσθετα στοιχεία, ένα τελείως άχρηστο γιατί έχει επικληθεί τόσες πολλές φορές πλέον που δεν ε, υπάρχει λόγος να επιμείνουμε επί της ανάγκης να υπάρχει αποτελεσματικό PNR και κατά δεύτερον μία πρόταση από τα συμπεράσματα του Φεβρουαρίου που καλεί τις μυστικές υπηρεσίες να έχουν μεγαλύτερες συνεργασίες. Αυτό το πράττουμε όχι μόνο από το Φεβρουάριο και, μετά, αλλά ιδιαίτερα μετά το Φεβρουάριο. Έχουν λοιπόν εντατικοποιηθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και η κοινή δουλειά, οι κοινέ επιχειρήσει. Για τα εξωτερικά σύνορα. Ο Ραούλ έχει πει τα πιο πολλά στοιχεία τα οποία μας ενδιαφέρουν. Αλλά θα ήθελα να πω το εξή. Πιστεύω ότι αποτελεί σημαντική βελτίωση να συμφιλειωθούν δύο κόσμοι οι οποίοι δεν συνεργάζονται δεν συνεργάζονταν επαρκώ. Έχουμε μια θεσμική χειροφένεια, αν θέλετε. Επί 15 χρόνια αναπτύσσουμε συστήματα διαχείρισης των συνόρων και τη μετανάστευση και ασύλου βάσει της νομικής ε, βάσης ε, της Ένωσης του πρώτου πυλώνα και σε άλλη συνθήκη με άλλη νομική βάση καταπολεμούμε την εγκληματικότητα και άρα είναι δύσκολο να υπάρξει συνεργασία των δύο αυτών στοιχείων και εκ παραλλήλου όλοι συμφωνούμε ότι στα σύνορα όλοι θα πρέπει να τα χειριζόμαστε και τις μεταναστατικές ροές και να φροντίζουμε για την ασφάλεια. Η Frontex δε όταν συλλέγει σχετικά στοιχεία στην ε, Μεσόγειο σε ό,τι αφορά και τους έτοντες άσυλο διαθέτει πάρα πολλές πληροφορίες που θα μας βοηθούσαν να είμαστε αποτελεσματικοί κατά του οργανωμένου κλίματος και της διακίνησης ανθρώπων. Οι υπουργοί ζητούν από τη Europol και τη Frontex από 1η Ιανουαρίου να ανταλλάσσουν πληροφορίες εφόσον το EDPS αποφανθεί έτσι. Οι υπουργοί λοιπόν συμφώνησαν να αναθέτουν ε, πιο πολλές αστυνομικές δυνάμεις από τις Europol στα hot spots προκειμένου να γίνουν πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι και έχουν συμφωνήσει ότι όσοι αντιμετωπίζουν μαζικές ε, μεταναστευτικές ροές, αν χρειαστεί θα πρέπει να λάβουν και τα απαραίτητα ηλεκτρονικά μέσα. Ε, συσκευές ανάγνωσης, διαβατηρίων, ηλεκτρονικές συσκευές, Europol και το καθεξής. Είναι σημαντικά λοιπόν όλα αυτά γιατί αυτά αποτελούν μια αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό φυσικά θα πρέπει να γίνει με πλήρη σεβασμό της νομικής βάσης. Δεν θέλουμε να μπλέξουμε διάφορες πολιτικές. Άσυλο και έγκλημα για παράδειγμα, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Η δεύτερη πτυχή. Τα υπόλοιπα τα εξήγησε, πολύ καλά ο Ραούλ για την ε, αντίδραση για την ποινική δικαιοσύνη. Θα γίνει και σχετική τροπολογία για την, το σχέδιο απόφαση για την τρομοκρατία για να ενταχθούν τα όσα προβλέπει και το ψήφισμα 2178 του ΟΗΕ. Αλλά έχουμε και άλλα στοιχεία. Καταρχάς, οι ψηφιακές, τα ψηφιακά αποτεκτικά στοιχεία. Καλό είναι να λέμε ότι θα στείλουμε όλου του κρατούμενου στη φυλακή, αλλά χωρί τα σχετικά αποτεκτικά στοιχεία δεν πρόκειται να το πετύχουμε αυτό. Δεν πρόκειται να καταδικαστούν. Στο πλαίσιο ενό κράτου δικαίου θα πρέπει να υπάρχουν αδιάστηστα αποτεκτικά στοιχεία. Αυτό είναι δύσκολο γιατί δεν συνεργαζόμαστε με τον Ασάντ ούτε είμαστε στη Συρία. Άρα θα πρέπει να συλλέγουμε τέτοια στοιχεία. Και τα μοναδικά πρακτικά στοιχεία είναι αυτά που πετυχαίνουμε από email, από παρακολούθηση τηλεφωνικών συνομιλιών και αυτό δεν είναι πολύ εύκολο γιατί τα πιο πολλά ψηφιακά στοιχεία έχουν αποθηκευτεί στις ΕΠΑ και θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε 8 μήνες στην καλύτερη περίπτωση. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο η Προεδρία έχει αρχίσει να αρχίσει να επενδύει προς την κατεύθυνση αυτή και η μελλοντική Ολλανδική Προεδρία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν και συζητήσεις και με τις ε, αρχές των ΗΠΑ. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο αναφέρθηκε και το οποίο για μένα αποτελεί σημαντικό στοιχείο είναι η αποκατάσταση Καλώς ορίζω την απόφαση της Επιτροπού Γιουρεβά με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, γιατί χρειαζόμαστε λοιπόν προγράμματα αποκατάστασης. Εδώ ε, δεν ε, είμαστε αρκετά ε, ενεργοί. Θα πρέπει να βρούμε επαρκείς λύσεις επανένταξης για τα άτομα αυτά, επαρκείς εναλλακτικές λύσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακόμα και αυτοί που θα πάνε τελικά φυλακή, δεν θα έχουν ένα πρόγραμμα για να ξεπεράσουν αυτή την ριζοσπαστικοποίηση στη φυλακή. Όχι, επιτείνονται τα φαινόμενα αυτά αντιθέτως. Και αυτό όχι μόνο προς το δικό του συμφέρον, αλλά προς το δικό μας συμφέρον βασικά. Κάτι άλλο. Και φαντάζομαι ότι η Λιβιέ θα αναφέρει τις σχετικές εξελίξεις στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά το δίκτυο ριζοσπαθικοποίηση, αριστεία 25 εκατομμυρίων. Αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία, αυτό το δίκτυο ριζοσπαθικοποίηση και όλο και πιο πολλά τρίτα κράτη μα ζητούν να τα βοηθήσουμε στο επίπεδο αυτό. Θα θέλαμε να υπάρχει μεγαλύτερη εξωτερική δραστηριότητα για να υποστηριχθούν τα κράτη-μέλη. Και το ίδιο ισχύει και για μια άλλη πρωτοβουλία που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συριακή ομάδα στρατηγικής επικοινωνίας. Αυτό είναι μια προσπάθεια που στέθηκε από επιτυχία και βοήθησε τουλάχιστον το ίμιση των κρατών μελών να σχεδιάσουν μια πιο στρατηγική μέθοδο επικοινωνίας σε μια προσπάθεια να ακουστούν ήπιες ε, φωνές στην κοινωνία των πολιτών να ακουστούν οι μετριοπαθείς. Ξέρουμε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να διαδοθεί αυτή η πρωτοβουλία. Το άλλο αφορά μια, ένα φόρουμ με την ιδανική κοινότητα. Γνωρίζω ότι ο Επίτροπος Αβρα, Αβραμόπουλος οργανώνει την Πέμπτη το απόγευμα μια συνάντηση με τις εταιρείε του διαδικτύου. Πιστεύω ότι είναι κομβική σημασία για να μπορέσει να υπάρχει μια συμφωνία ε, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να διαγράφονται τα παράνομα, οι παράνομες ιστοσελίδες. Αλλά βεβαίως καλούμεθα να κάνουμε πολύ περισσότερα. Αν θυμάστε τη δήλωση του Φεβρουαρίου, είπαμε, κάναμε μία αναφορά στον εξτρεμισμό ε, σε πολλούς τομείς, ε, στον τομέα της εργασίας, ε, του πολιτισμού. Και αυτό είναι κάτι που απασχολεί την Επιτροπή. Σίγουρα θα εκδοθεί, ένα ανακοινωθέν από, τον αρμόδιο επίτροπο. Εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχουν προγράμματα, να βαρχίδες θα λέγαμε, να θυμηθούμε τι έκανε ο πρόεδρος ε, Ομπάμα όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα εικονικής ανταλλαγής. Χρησιμοποίησε το ίντερνετ για να διασυνδεθούν ένα εκατομμύριο Αμερικανοί με ένα εκατομμύριο Άραβες για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο ίδιος καθηγητής ε, διδάσκει τα ίδια ε, μαθήματα και πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πώς αυτό είναι ικανό να άρει τα στερεότυπα στους νέους, ε, στους ε, εφήβους. Αρέσει πάρα πολύ το ίντερνετ και το διαδίκτυο θα μπορούσε να είναι μια πραγματική γέφυρα. Ο, είπατος, ε, ε είπατε η εκόραση είναι και εγώ, καταβάλουμε προσπάθειες να ενθαρρύνουμε συνεργασία σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας με τις χώρες της Μεσογείου. Ε, πρόσφατα συνεργαστήκαμε με την Τινησία. Αυτή είναι μια νέα προσέγγιση. Θέλουμε να συνεργαστούμε από κοινού, να κινητοποιήσουμε τα οικονομικά προγράμματα για να ενδυναμωθεί η δυνατότητα αυτών των χωρών να αντιμετωπίσουν τις άπειρες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες. Κάναμε το ίδιο με την Ιορδανία, με την Τουρκία, με το Μαρόκο, με όλες τις χώρες της Μεσογείου αναπτύξα, ε, ε, τοποθετήσαμε έναν επιτετραμένο για θέματα αντιτρομοκρατίας αυτές τις χώρες. Μας απασχολεί το θέμα της ασφάλειας των πτήσεων, το θέμα της χρηματοδότησης ε, του, της τρομοκρατίας κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Κερχόβα. Ο κύριος Λάξ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, δεν θέλω να επαναλάβω όλα τα σημαντικά που είπαν οι συναδελφοί μου στις προηγούμενες παρουσιάσεις τους, να δώσω ορισμένα περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειε για τα όσα έχουμε προτείνει και θα προτείνουμε με τι επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Ο Ζιλ ανέφερε το κέντρο αριστείας, το οποίο είναι πλέον επιχειρησιακό από τον Οκτώβριο και θα επεκταθεί, θα λάβει περισσότερη χρηματοδότηση, περισσότερο προσωπικό και θα έχει και νέε ομάδες εργασίας. Μεταξύ άλλων και μία για την εκπαίδευση, μία ε, για τις ε, οικογένειε και κοινότητες για να αντιμετωπίσουμε τα πρώτα σημάδια της ριζοσπαστικοποίηση και την άμεση ανταπόκριση ως προς αυτήν την ριζοσπαστικοποίηση γιατί όπως αναφέρθηκε η φυλάξη δεν είναι η πανάκια. Πράγματι θα ξεκινήσει και το IT Forum την Πέμπτη Σκοπός είναι να υπάρξει ένας διαθετικός διάλογος ε, και με τον ε, κλάδο της τεχνολογίας για να έχουμε και τις γνώσεις τους, τη στήριξή τους ό,τι αφορά το τεχνολογικό σκέλος αλλά και πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ε, αυτή την αντίθετη, το αντίθετο αφήγημα αν θέλετε πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε ακριβώς αυτή τη διαδικασία ρυθμιστικοποίησης από τις κοινότητες και για τις κοινότητες. βλέπουμε ότι είναι κάτι το οποίο τους ενδιαφέρει ιδιαίτερο και θα θέλαμε ε, να συμφωνήσουμε επί ορισμένων συγκεκριμένων ενεργειών. Ελπίζουμε να ξεκινήσει μια φάση 2 της ε, στρατηγικής ομάδας ε, συνεργασίας, SCAT. αυτό βεβαίως είναι, πρόκειται για πυρογνώμονες τηλεπικοινωνιών και επικοινωνίας, όχι μυστικών υπηρεσιών που βοηθούν κυβερνήσεις και τοπικούς φορείς να καθορίσουν ε, την πολιτική επικοινωνία τους. Τώρα, για τα όσα συμφωνήθηκαν την ε, προηγούμενη εβδομάδα. Δυστυχώς τα πυροβόλα όπλα και ιδίω ε, τα πολυβόλα όπλα και οι εκρητικές ύλες μάλλον θα εξακολουθήσουν να είναι το ε, μέσο που θα προτιμούν οι τρομοκράτες. Γιατί είναι εύκολο κάποιος να έχει πρόσβαση σε αυτά και είναι και πιο εύκολα στη χρήση τους ε, σε σχέση με άλλα μέσα. Γι' αυτό και την περασμένη εβδομάδα προτείναμε έναν αυτόνομο κανονισμό της Επιτροπής που θα εναρμονίζει τα πρότυπα για την ε, απενεργοποίηση των πυροβόλων όπλων γιατί δεν ισχύουν τα ίδια τεχνικά πρότυπα σε όλα τα κράτη-μέλη. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να αγοράσει ένα παροπλισμένο Καλάσνικοφ ή M16 ή οποιοδήποτε άλλο περιβολόπλο και είναι εύκολο να το επανεργοποιήσει. Τώρα λοιπόν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτό και όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν τα ίδια τεχνικά πρότυπα. Ούτω ώστε όταν ένα ε, στρατιωτικό πυροβόλο όπλο έχει παροπλιστεί, αυτό να είναι μόνιμο άπαξ και διαπαντός. Και το δεύτερο μέσο είναι μία οδηγία που επανεξετάζει ή μάλλον μέχρι τώρα η ισχύουσα νομοθεσία αφορούσε ε, την παραγωγή, θέση εμπορία ε, και διακίνηση των ε, όπλων αυτών που αφορούσαν όμως περισσότερο κυνηγητικά όπλα και το καθεξής. Υπήρχε λοιπόν μια σημαντική πτυχή ως προς την εσωτερική αγορά. Τώρα εμείς έχουμε εισαγάγει και μία ε, πολύ ισχυρή ε, παράμετρο ασφαλείας. Θα δείτε και την οδηγία εν το χρόνο, όμως ε, θέλουμε να υπάρχει ουσιαστικά πολύ πιο ε, ουσιαστικός έλεγχος σε άδειε αγοράς όπλων. Για τα στρατιωτικά πυροβολά όπλα βεβαίως αυτά θα απαγορεύονται εντελώς, αλλά και για τα κυνηγητικά όπλα, γιατί κάποια είναι εξίσου ή και πιο ισχυρά από τα καλάσνικοφ σε ό,τι αφορά το διαμέτρημα και το καθεξής. Αν πάει κάποιος στην Αφρική και θέλει ε, να σκοτώσει ένα βουβάλι, για παράδειγμα, δεν ισχύει σε δική μου περίπτωση, αλλά μπορεί κάποιος να αγοράσει ένα κυνηγετικό όπλο το οποίο είναι πιο ισχυρό από τα υπόλοιπα. Και μπορούν να πάρουν και τη μορφή του ημιαυτόματου πολύ εύκολα. Όλα αυτά πρέπει να τα εκτάσουμε με προσοχή λοιπόν. Αύριο, αν όλα πάνε Κατευχήν, η Επιτροπή θα υιοθετήσει ένα νέο σχέδιο ενεργειών και δράση και για τις δύο κατηγορίες όπλων. Θα έχουμε και νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα για το ίδιο ακριβώ ζήτημα. Για να υπάρχει καλύτερη συνελασιμότητα, έλεγχος, ζητήματα μαύρη, αγοράς και φαιών ζωνών. Τι εννοούμε με τι ζώνες ε, ορισμένα παζάρια για παράδειγμα με ε, όπλα αντίκες ε, για συλλέκτες. Σε αυτά λοιπόν ε, θέλουμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ζώνες, να απαγορεύσουμε και να επαρεμποδίσουμε την πώληση όπλων αλλά και εξαρτημάτων στο διαδίκτυο. Θα μπορεί κάποιος να κάνει την παραγγελία, αλλά μετά θα πρέπει αυτοπροσώπως να πάει κάποιος και να παραλάβει το θέμα. Σε ό,τι αφορά τι εκρητικές ύλε, τώρα, οι έρευνες δείχνουν ότι η εκδική ύλη που χρησιμοποιήθηκε ε, στο Παρίσι είχε ε, παραχθεί από πρόδρομες ουσίες που είναι εύκολο κανείς να τις αγοράσει. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μάλλον η πρόταση που υιοθετήσαμε πέρσι το 2014 φαίνεται ότι δεν έχει εφαρμοστεί πλήρω για τις πρόδρομες ουσίες. Τα κράτη-μέλη δηλαδή δεν έχουν κάνει τα απαραίτητα. Θα υπάρξει και αναθεώρηση βεβαίως το 2017 θα υποβάλουμε την πρόταση αναθεώρηση για να έχουμε πιο στενού ελέγχους και απαγορεύσει, αλλά να προσθέσουμε και νέες ουσίε σε αυτές τις απαγορευμένες πρόδρομες ουσίε που μπορεί κάποιο ε, να παρμηθευτεί από τον τομέα των καλλιτικών, τη κυπουρική ε, και το καθεξή. Τώρα για την οδηγία. Πράγματι αύριο, αν όλα πάνε βάσει σχεδίου, η Κομισιόν θα υιοθετήσει μια νέα νομοθετική πράξη που όχι μόνο θα τροποποιήσει την υφιστάμενη απόφαση πλαίσιο ε, ε, σε ευθυγράμμιση και με ε, το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα έχουμε όμως μία οδηγία που θα συγκεντρώνει όλο το κεκτημένο σε ό,τι φορά την ποινικοποίηση αυτών των αδικημάτων. Βεβαίω θα βασιζόμαστε στους υφιστάμενους ορισμούς το 2002, όπως έχουν τροποποιηθεί το 2008 και θα έχουμε και τα δικήματα που συνδέονται με τους αλλοδαπούς μαχητές, όπως είναι ε, το ταξίδι για τρομοκρατικού σκοπούς, ε, παθητική κατάρτιση, χρηματοδότηση τέτοιων ε, δρομολογίων και ούτω καθεξής. Θα δείτε λοιπόν ε, το κείμενο σύντομα και θα υιοθετηθεί αύριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα άλλο καθήκον που έχουμε αναλάβει από τους υπουργούς. Τι μπορούμε να κάνουμε. Το ότι FTB ανέφερε ο συνάδελφος. Πράγματι, αυτές οι πληροφορίες ε, τροφοδοτούν ε, τις συνεχιζόμενες έρευνες και στη Γαλλία και στο Βέλγιο και είναι εκατοντάδες τα στοιχεία Επομένω, ε, φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικό μέσο. Όμω δεν αρκεί. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια χαρτογράφηση όλων ε, των ε, οικονομικών μέσων που έχουμε ή δεν έχουμε στη διάθεσή μας και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Και εδώ αναφέρομαι και όλα αυτά είναι ερωτηματικά βεβαίως. Μήπως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τους κανονισμούς ροών ρευστού. Τι πρέπει να κάνουμε για τα εικονικά νομίσματα, τα ψηφιακά νομίσματα και τα bitcoins. Θα πρέπει να ποινικοποιήσουμε το ξέπλυμα μαύρου χρήματο. Υπήρξε στην απόφαση πέρσι για την τέταρτη οδηγία κατά του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Όμως, δεν έχει αναγνωριστεί ως ποινικό αδίκημα το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μήπως θα πρέπει να γίνει αυτό. Μήπω επίση θα πρέπει να βάλουμε πρόταση για το άρθρο 75 της συνθήκης για να περάσουμε σε δίμευση περιουσιακών στοιχείων όταν έχει αναγνωριστεί μια τρομοκρατική οργάνωση. Θα πρέπει αυτό να αναπόκειται στα κράτη-μέλη. Κάποιοι έχουν ε, ε, ένα συγκεκριμένο σύστημα, άλλοι δεν έχουν τίποτα για το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων. Γιατί μέχρι να περάσουμε στη διαδικασία των κατασχέσεων και τα καθεξής έχουν φύγει όλα αυτά τα χρήματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς αυτό θα γίνει με αναλογικό τρόπο, να μην επηρεάζουν τα κρατημέλη που ήδη έχουν αντίστοιχο σύστημα και να συνάδει και με το αντίστοιχο σύστημα του ΟΗΕ. Εδώ λοιπόν υπάρχει προσταθημένη αξία, όμως αυτή τη στιγμή μας έχουν ζητήσει να κάνουμε μια, ένα εγχείρημα χαρτογράφησης για τις μελλοντικές μας εργασίες. Κλείνοντας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι αν όλα πάνε βάσει σχεδίου θα υιοθετήσει στις 15 Δεκεμβρίου ε, το πακέτο για τα ευφυή e e σύνορα. Και θα εξετάσουμε μια στοχοθετημένη τροποποίηση του συστήματος SIS, του σύστημα πληροφόρησης Schengen. Αντίστοιχα, ε, θα επεταχύνουμε και ε, θα τροποποιήσουμε και το σύστημα έκρης για τις ε, ποινικέ πληροφορίε που δεν χρησιμοποιείται επαρκώς, αφορά την ανταλλαγή ποινικών μητρών, ιδίω για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Εάν δηλαδή έχουμε κάποιον που έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για ένα ποινικό αδίκημα και δεν το γνωρίζουμε, αυτό είναι μια κρίσιμη σημασία πληροφορία. Πρέπει να την ξέρουμε σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών ε, πέραν των όσων είπε ο Τζιλ, έχουμε και την απόφαση Προύμ που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη και τις αρχές επιβολής του νόμου αλλά και τις αρχές ασφαλείας να ανταλλάσσουν δεδομένα DNA, ε, δακτυλικών αποτυπωμάτων και αδειών κυκλοφορίας. Δεν αξιοποιείται. Δείτε τι έγινε στο Παρίσι. Αυτές οι τρεις κατηγορίες πληροφοριών θα ήταν αποφασιστική σημασία για να εμποδίσουμε τους δράστες από το να φτάσουν και να φύγουν από τον χώρο της επίθεσης. Υπάρχει, αλλά δεν αξιοποιείται στο έπακρο. Θα το εξετάσουμε. Τέλος. Έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα και συμφωνώ, αλλά με μια ε, μικρή μνήα υπάρχει μια σημαντική ε, μεταβολή στο φόρο του Σεπεράντη ε, σε αυτές τις τρομοκρατικές ομάδες σε σχέση με ορισμένες ε, δεκαετίες. Παλιότερα, λοιπόν πριν από μερικές δεκαετίες, στοχοθετούσαν πολιτικούς στόχους. Τώρα όμως έχουμε αυτούς τους soft targets. Πάνε σε μαραθώνιους, σε μουσεία, σε πλατείες, σε θεατόρια, σε θέατρα. Ξέρουμε ότι την περασμένη φορά έλαβαν οδηγίες από τους ε, επικεφαλείς τους ε, στη Συρία και στο Ιράκ. Εάν δεν μπορούν να πάνε στο Χαλιφάτο, να κάνουν αυτόν τον τζιχάντ όπου και αν βρίσκονται και με όποιο τρόπο έχουν στη διάθεσή του, Με μαχαίρι, με όπλο, με ό,τι έχουν στα χέρια τους. Και ξέρουμε ότι αυτή η οδηγία έχει μεταδοθεί μέσω των μηχανισμών προγάντας τους. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν είμαστε σε στενή συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες των κρατών μελών για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ακριβώς για να δούμε πώς ε, μπορούμε να διασφαλίσουμε τους soft targets όπως είναι ε, τα αεροδρόμια, όπως είναι ε, οι δημόσιες εκδηλώσεις. Έχουμε κάνει ορισμένες δοκιμές και θέλουμε να έχουμε και ένα εγχειρίδιο για του για τις αρμόδιες γιατί και οι πόροι είναι περιορισμένοι στην αστυνομία, για παράδειγμα. Πρέπει να δούμε πώ θα μεγιστοποιήσουμε την αποδοτικότητα των δυνάμεών μα, χωρί να υπάρξει απαραίτητα αύξηση χρηματοδότηση, να καταφέρουμε να προστατεύσουμε περισσότερο ε, τους ε, στόχους μας. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ και τους τρεις. Ε, θίξατε πολλά ζητήματα. Έχουμε και έναν πλήρη κατάλογο μελητών. Προηγουμένω αναφερθήκατε και στην απόφαση του ΦΥΜ που ελήφθη το 2005 για την ανταλλαγή δεδομένων DNA, των αποτυπωμάτων και αδειών κυκλοφορία. Δεν υπάρχει επαρκή ανταλλαγή στα, στα περισσότερα κράτη-μέλη. Αυτό θα είχε βοηθήσει βεβαίω την αντιμετώπιση των μικροτικών επιθέσεων. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα ε, μη επαρκούς λειτουργίας των κυβερνητικών συμφωνιών. Είναι ένα ζήτημα υλοποίησης αλλά και νέα νομοθεσία και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει με θετικό πνεύμα βέβαια στην Επιτροπή μας. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν κάποια κέρια ζητήματα μη υλοποίηση νομοθεσία ε, που σίγουρα θα θίξουν και οι συνάδελφοι. Κυρία Χόλμαγερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις πολύ, για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Έχω τόσες πολλές ερωτήσεις και φαντάζομαι το ίδιο θα έχουν και οι συνάδελφοι για το θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Είναι θέμα αδράνειας αυτό, αυτή είναι η αιτία για το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη και οι αστυνομικές και μυστικές τους υπηρεσίες δεν ανταλλάσσουν πληροφορίας. Είναι αμέλεια. Υπάρχουν δυσκολίες στα κράτη-μέλη μήπως σε ό,τι αφορά τη συλλογή των σχετικών ε, δεδομένων και την ανάλυση τους θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι αιτίε, τι οδηγεί σε αυτή την ελλειπή συγκέντρωση δεδομένων. Κάποιοι πιστεύουν ότι φταίει και η προστασία των δεδομένων ε, για την ελλειπή ανταλλαγή τέτοιων στοιχείων. Αν αυτό ισχύει, πείτε μας επακριβώς τι παρουσιάζει πρόβλημα και ποια είναι τα προβλήματα. Ακούσαμε και για, ε, για το Eurodac ότι δεν είναι δυνατή η αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων, αλλά αν σωστά καταλαβαίνω η Frontex έχει ως στόχο μια τέτοια μορφή ανταλλαγή δεδομένων. Θα ήθελα πιο πολλές πληροφορίες, γιατί τουλάχιστον άμα υπάρχουν προβλήματα να τα ξέρουμε εδώ στο Κοινοβούλιο, να κάτσουμε να τα συζητήσουμε. Στη συνέχεια, άλλη μια ερώτηση έχω να κάνω για την συνεργασία με την, Ισία, την Ιορδανία και την Τουρκία αλλά και με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμπεριληφθούν και κάποιες αξιόπινες ποινικέ πράξεις στα δεδομένα αυτά. Πώς θα διαμορφωθεί ακριβώς αυτή η τελαγή δεδομένων και άμα συμπεριληφθούν τα ποινικά αυτά στοιχεία. Το πρόβλημα της Τουρκίας προβλέπει, για παράδειγμα, η Τουρκία ε, ποινικό έγκλημα, για παράδειγμα την ε, έκφραση λόγου, την ε, απαγόρευση διαδήλωσης. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη διαφορά, αν πρόκειται για σοβαρές εγκληματικές πράξεις, όπως για παράδειγμα δολοφονία κτλ. Ή περιλαμβάνονται όλες αυτές οι αξιόπινες πράξεις και πώς θα διαμορφωθεί λοιπόν αυτή η συνεργασία. Και τελευταία, ερώτηση για τις εκρηκτικές ύλες. Συχνά έχουμε συζητήσει το γεγονός ότι για παράδειγμα στα ναρκωτικά όπως και στα εκρηκτικά θα πρέπει να υπάρχει πιο μεγάλη υποχρέωση καταχώρησης και αυτό θα πρέπει να οδηγεί σε άρα άραγε των υλών αυτών. Ποια είναι η κατεύθυνση της νέας αυτής ε, ρύθμισης. Ευχαριστώ κυρία Σίπελ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ έχω πολλέ ερωτήσει και πολλέ παρατηρήσει να κάνω, αλλά θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ σε κάποια θέματα. Καταρχά, αφού το ακούσαμε και του τρει ομιλητέ, κατανοούμε ότι πλέον υπάρχει μία συμφωνία ότι η αντιμετώπιση των θεμάτων σε εθνικό και μόνο επίπεδο δεν επαρκεί. Και αυτό αφορά τα θέματα ασφάλειας και τα κρατημέλη θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι εθνικές λύσεις στις σημερινές προκλήσεις δεν αρκούν. Αλλά επιμένουν στο θέμα της εθνικής κυριαρχίας. Διάβασα μια συνέντευξη του 2012 του Helmut Schmidt, του πρώην καγκελάριου, που ανέφερε ότι δεν υπάρχει πλέον εθνική κυριαρχία γιατί μας δεσμεύουν πολλές, ε, πολλές διεθνείς συμφωνίες και συνεργαζόμαστε με άλλα κράτη και οι προκλήσεις είναι υπερβολικά μεγάλες για να αντιτηρήσουμε επικυριαρχίες εθνικές. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν το συνειδητοποιούμε αυτό και έχω διάφορα παράδειγματα να σας πω από το εσωτερικό της Γερμανίας για ελληπή ανταλλαγή ε, δεδομένων μεταξύ των υπηρεσιών της Γερμανίας. Πώς θα βελτιώσουμε λοιπόν την κατάσταση. Υπάρχουν εργαλεία διάφορα είδη εργαλείων, αλλά δεν αξιοποιούνται. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, πιστεύω, και αυτό ενδεχομένως να αποτελέσει και το πρόβλημα για το μελλοντικό PNR, γιατί το αναφέρουμε ως ευρωπαϊκό PNR, αλλά ουσιαστικά θα είναι 29 διαφορετικά συστήματα, η ευρωπαϊκή οδηγία και τα 28 εθνικά συστήματα, όπου οι εθνικές αρχές θα αποφασίσουν επί των κριτηρίων και όσο σήμερα δεν είναι σίγουρο κατά πόσον θα είναι υποχρεωτική πραγματικά η ανταλλαγή δεδομένων για τη χρήση των υφιστάμενων εργαλείων. Θα ήθελα να ανακαλύψουμε το τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου τα στοιχεία που προέρχονται από τα κρατημένη. Έχουμε το σύστημα σε Σέγγεν, το ΑΠΗ, την κοινή ερευνητική ομάδα Με τις τρομοκρατικές επιθέσεις λοιπόν στην Ευρώπη, αν ρωτιέμαι γιατί είναι τόσο απλό να αγοράσει κανείς όπλα στην Ευρώπη, έρχονται λοιπόν ε, στην Ευρώπη, μπορεί κανείς να αγοράσει ε, τέτοια όπλα σε σταθμούς ε, και τα ξέρουν αυτά οι τρομοκράτες, είναι γνωστά. Μου λένε καμιά φορά, μα δεν ξέρεις ότι μπορεί να αγοράσεις όπλα σε αυτόν τον σταθμό. Εμά όχι, δεν το ήξερα και ούτε η αστυνομία φαίνεται ότι το ήξερε, αλλιώ θα είχε κάνει ελέγχου. Εδώ υπάρχει λοιπόν πρόβλημα για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Σύμφωνο ότι αυτό αποτελεί κοινό ευρωπαϊκό καθήκον. Όσο μιλάμε για τον έλεγχο των συνόρων μα, όχι για το κλείσιμο των συνόρων μα για του μετανάστε. τι σημαίνει όμω αυτό να λέμε ότι είναι κοινό ευρωπαϊκό καθήκον. Ω τώρα δεν βλέπω τα κράτη-μέλη μας να είναι έτοιμα. Να πούν ότι εντάξει, κοιτάξτε, θα σας δώσουμε τις τεχνικές δυνατότητες, τη χρηματοδότηση για να διασφαλίσουμε ότι τα εξωτερικά σύνορα ελέγχονται επαρκώς. Δεν μπορώ, θεωρώ, δεν μπορούμε, ε, θεωρώ, να το αφήσουμε αυτό στα χέρια των ε, κρατών μελών που έχουν εξωτερικά σύνορα. Είναι κοινό ευρωπαϊκό καθήκον. Και ανησυχώ γιατί τα κράτη-μέλη δεν έδειξαν αρκετά χρήματα στην ε, υποτερμοστία του ΟΗΕ, στο αφρικανικό καταπίστευμα, να δούμε τι θα γίνει με την Τουρκία τώρα. Θα δώσουν λοιπόν στη τελική ανάλυση τίποτα για να εκπληρωθούν αυτές οι υποχρεώσεις για τον έλεγχο των συνόρων. Δεν είμαι καθόλου βέβαιη για την ε, περιοχή Σέγγεν και τον έλεγχο των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει να σας πω ότι ανησυχώ ανησυχώ γιατί αναρωτιέμαι είναι απαραίτητο, θα ήταν απαραίτητο αν όλα τα υπόλοιπα εργαλεία λειτουργούσαν άψογα σε ό,τι αφορά την πρόληψη, την ε, αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίηση, την απάντηση σε τέτοια μηνύματα, όλα αυτά ναι, είναι απαραίτητα και πραγματικά ελπίζω, ελπίζω λέω ότι θα εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή με συνέπεια και με επιμονή, όχι τώρα μετά τις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις και ίσως και πριν από κάποιες μελλοντικές τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά ότι δεν θα περιοριστούμε μόνο σε θέματα ασφάλειας, αλλά και για να κάνουμε τους πολίτες μας να αισθανθούν μέλη αυτής της κοινωνίας, όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, αλλά και στην γενικότερη κοινωνία. Η κυρία Στίβενς. Thank Ο κύριος Στίβενς. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος ε, της ΙΣΙΑΣ ό,τι αφορά την ανάγκη για τις χώρες μέρη να θέσουμε ως προτεραιότητα τα μέσα εφαρμογής. Βεβαίω χρειαζόμαστε περισσότερα μέσα στη διάθεσή μας, αλλά θα πρέπει να συμβάλλουμε έτσι ώστε να λειτουργήσει καλύτερα αυτό που ήδη έχουμε. Δηλαδή, να είναι βασική προτεραιότητα η ανταλλαγή ε, Πρωτιβολιών. Το θέμα είναι να αντιμετωπίσουμε την ριζοστικοποίηση. Οι χώρες μέλη θα πρέπει να κάνουν κάτι περισσότερο από όσα αναφέρατε. Θα υπάρξει μία πρόταση για ε, συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ή FTP για το πρόγραμμα οικονομικού εντοπισμού τρομοκρατών. Είναι κάτι που θέλουν οι χώρες μέλη. Μιλάμε για την ανάγκη ισχυρο, ισχυρότερου ή αποτελεσματικότερο κότερου ελέγχου στα σύνορα. Τι περιμένουμε να υποβληθεί μια άλλη πρόταση, τι κάνει η Frontex. Εξ ονόματο ε, της αντιπροσωπεία NBA θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει προστιθέμενη αξία στην καταπολέμηση τη τρομοκρατίας ε, λόγω του διακρατικού τρόπου λειτουργία των δραστών. Οι Ευρωπαίοι πολίτε αναρωτιούνται γιατί δεν έχει γίνει, δεν έχει επιτευχθεί πρόοδο μετά στι επιθέσει. Πάρτε για παράδειγμα το ENU, PNR, το φάκελο αυτό, ο οποίος ε, ε, έχει σταματήσει λόγω της παρακόλλησης από πλευράς του κυρίου Βερχόφτατα. Πολύ συχνά κατηγορούνται οι υπηρεσίες πληροφοριών. Δεν χρειάζεται να κατηγορήσουμε τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει σχέση με εμά τους ίδιους. Συνεπώς θα επιθυμούσα για μία ακόμα φορά να ζητήσω από όλους σας να βάλετε κατά μέρος τους δογματισμούς σας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα σενάρια καταστροφής που θα επακολουθήσουν. Βεβαίω θα πρέπει να επιτευχθεί μια ισορροπία, αλλά πραγματικά και με τρόπο απελπιστικό χρειαζόμαστε ε, και πρόοδο. Κυρία Βίνστρομ. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό. Ε, ε, με μεγάλο ενδιαφέρον ακούω τους συναδέλφους θα ε, ήθελα να κάνω μία ερώτηση στην Επιτροπή σχετικά με την ε, πρόταση ελέγχου που γίνεται. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν πάρα πολλοί μαχητές, πολλοί υπάρχουν στην Σουηδία και στην ίδια μου τη χώρα υπάρχουν, α, με συγχωρείτε, υπάρχουν πάρα πολλοί κυνηγοί οι οποίοι νόμιμα χρησιμοποιούν όπλα και αυτό γίνεται παντού. Τις τελευταίες εβδομάδες έλαβα έναν αριθμό πολλές, πολλές ερωτήσεις, ε, πολλές επιστολές που μου έλεγαν εξετάστε το θέμα των Σουηδών κυνηγών. Ε, αυτή είναι πολίτες νομοταγείς που χρησιμοποιούν τα όπλα. Η πρόταση αυτή δεν θα αντιμετωπίσει σοβαρότατα θέματα όπως το θέμα των παράνομων όπλων που εισέρχεται από πολλά, πολλές μεριές στις χώρες μας. Το ερώτημά μου είναι τι θα θέλατε να πω εγώ στους πολίτες. Μπορούμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι η πρόταση της Επιτροπής θα είναι αναλογική και αποτελεσματική και ότι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα παράνομα όπλα και να αφήσει ήσυχους τους κυνηγούς να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Okay, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αργεντίνη. Εμένα δεν με απασχολούν τόσο πολύ οι κυνηγοί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και η Αντρομοκρατική ε, ομάδα μιλάνε πάρα πολύ για τον έλεγχο των συνόρων για αυτού που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν κοιτάξουμε όμω τι επιθέσει που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, προήλθαν από ανθρώπου που ήταν πολίτε αυτών των χωρών. Το θέμα είναι τι ε, θα κάνουμε όταν οι ε, γονείς ακούνε ότι το παιδί τους θα φύγει για να πάει στη Συρία και τι θα γίνει και με τη μετανάστευση. Ε, το, το γνωρίζουμε όλα αυτά. Θα ήθελα να συζητήσουμε λοιπόν αυτό το, αυτή την εκροή. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι τα νεαρά παιδιά, οι νεαροί άντρες και γυναίκες δεν θα στραφούν προς τον εξτρεμισμό. Και δεν θα φύγουν για να κάνουν κακό κάπου αλλού. Ναι, έρχονται και πάλι εδώ λοιπόν για κακό, αλλά θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί την οδηγία κατά του ξεπλήματο χρήματο. Τον Ιούλιο νομίζω δημοσιεύτηκε. Είμαι εισηγήτρια για το θέμα αυτό. Το διαπραγματευτήκαμε μέχρι πέρσι τα Χριστούγεννα, δημοσιεύτηκε τελικά τον Ιούλιο. Και θα ήθελα πραγματικά πιο πολλέ πληροφορίε. Πού πιστεύετε ότι υπάρχουν κενά και τι θα κάνουμε για το γεγονός ότι το 2017 υποχρεούνται μόνο τα κρατημέλη να εφαρμόσουν την νομοθεσία αυτή. Και επίσης υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι τρομοκράτε στα δυτικά κράτη, κράτη είναι πολύ φθηνή η δράση τους. Ε. Πού ε, δαπανώνται πολλοί πόροι για τρομοκρατία στη Συρία. Αυτό λοιπόν πώς το αντιμετωπίζουμε. Αυτό έχει νόημα για τις ε, ψεύτικες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και θα ήθελα να καταλάβω το τι μας λείπει από αυτή την οδηγία κατά του ξεπλήματος χρήματος υπαρχών 4. Ποια κράτη-μέλη δεν έχουν κάνει περικοπές στις αστυνομικές δυνάμεις και στις περιπολίες ε, τα τελευταία χρόνια. Ούτε η Γαλλία, ούτε η Ιταλία, ούτε δική μου χώρα. Όλοι μειώσαμε τις δαπάνες για τις αστυνομικές περιπολίες. Και τώρα μας αναφέρουν οι ειδικοί για θέματα τρομοκρατίας την ανάγκη για καλύτερες θέσεις εργασίας και καλύτερες εκπαιδεύσεις. Και πραγματικά με προβληματίζει αυτό. Ξέρουμε τι χρειάζεται, αλλά δεν το κάνουμε αυτό. Γιατί? Αυτό ισχύει και για το κέντρο RAN, το δίκτυο ευαισθητοποίησης για την ριζοσπαστικοποίηση. Από τον Οκτώβριο έχει ξεκινήσει, αλλά δεν είναι αποτελεσματικό γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση και δεν ξέρουμε και δεν μπορούσαμε να αποφασίσουμε σε ποιον θα δώσουμε το συμβόλαιο. Αυτό πραγματικά αποτελεί ντροπή. Τέλος, μετά τη Ρήγα, Πρόεδρε, όλος ο κόσμος έκανε υποσχέσεις και τελικά δεν έγινε τίποτα. Το μήνυμα λοιπόν που μας ε, δίνουν είναι σας παρακαλούμε να είσαστε γρήγοροι για την εφαρμογή του PNR για να καταπολεμήσουμε τους τρομοκράτες. Μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτό το μήνυμα και να πούμε ότι κοιτάξτε, κάντε και εσείς αυτά που έχετε υποσχεθεί και φροντίστε τους Ευρωπαίους πολίτες και καταρχάς τις εκροές. Ευχαριστώ. Η κυρία Ινφέλτ. Ευχαριστώ. Πρώτα θα ήθελα να απαντήσω στον συνάδελφο και να αναφέρω ότι δεν ε, παρεμποδίζει κανένα τίποτα. Υπάρχουν διαπραγματεύσει στο PNR και εγώ διαπραγματεύομαι εξ ονόματο του Άλντε και δεν εκτιμώ το ότι φέρνετε τη βελγική πολιτική σκηνή ε, σε όλη αυτή τη συζήτηση και δεν λέτε την αλήθεια. Και θα περίμενα κάτι καλύτερο από εσά για να είμαι ειλικρινή σταματήστε να ψεύδεστε. Είναι ψέμα ότι το Κοινοβούλιο μπλοκάρει το PNR. Τελεία και παύλα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εισαγωγή σχεδόν μία ώρα ακούσαμε τους ομιλητές και μου είναι πάντα περίεργο γιατί ποτέ δεν ξέρω ποιος ακριβώς μας μιλά, μας απευθύνει τον λόγο. Εντάξει, η Προεδρία του Λουξεμβούργου αλλά ο κύριο Κέρκοβε επίση, μιλάει εξ ονόματο του Συμβουλίου. ποιο είναι ο συνομιλητή μα, Είναι περίεργη διαδικασία. Και επίση με προβληματίζουν δηλώσει του κυρίου Ντεκέρκοβ στα μέσα, όπου ουσιαστικά εμέσως ε, κατηγορεί το Κοινοβούλιο, την μπλοκάρει την απόφαση και, και τη λήψη αποφάσεων, ιδίω για το PNR. Όταν μιλούμε για την υπεράσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων κράτους δικαίου και δημοκρατικών ελευθεριών, καλό θα ήταν να δείχνουμε και λίγο σεβασμό προς την κοινοβουλευτική δημοκρατία, κύριε Ντεκέρκχοβε. Έχω πολλά ερωτήματα. Θα ξεκινήσω από το PNR. Είναι ενδιαφέρον που κάποιοι λένε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, ε, το ανόητο κοινοβούλιο που μπλοκάρει όλες αυτές τις προτάσεις. Να πω κάτι που είπα και χθες. Η η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας ζωής και τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι πραγματικά θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν είναι ε, απλώς ε, σκέψεις κάποιων ε, αριστερών. Είναι θεμελιώδες δικαι... Ε, ελευθερίες που έχουν εγγραφεί ε, στο κράτος δικαίου. Η ομάδα μου, η Άλντε, κυρία Στέβενς, είχε προτείνει αρχικά να υιοθετήσουμε κανονισμό για το PNR και όχι οδηγία. Γιατί η οδηγία πρέπει να εφαρμοστεί και από τα 28 κράτη-μέλη και αυτό θα πάρει χρόνια. Ενώ ο κανονισμό εφαρμόζεται άμεσα. Και όπω είπαν και όλοι, είναι ιδιαίτερα επίγον. Γιατί δεν υπήρξε λοιπόν πλειοψηφία. Θα είχαμε γλιτώσει πολύ χρόνο. Αλλά νομίζω ότι ήσασταν αντίθετοι. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν. Επίση, η Βρετανία του Λουξεμβούργου θα μπορούσε να μα πει και να μα δώσει λίγη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τι μεμονωμένε επιμέρου θέσει των κρατών μελών στο Συμβούλιο, γιατί είναι ιδιαίτερα διαφανή τα πράγματα. Ξέρω ότι υπάρχει ε, διαφωνία ε, απόψεων σε πολλά ζητήματα, αλλά θα ήταν δίκαιο προ του πολιτέ στο Συμβούλιο να είναι ανοιχτό. Ποιο, τι θέση παίρνει ο καθένα. Αυτό το χρωστάτε και στο Κοινοβούλιο, αλλά και στου πολίτε. Εκτό και αν βεβαίω δεν θέλετε να είστε διαφανεί σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς ασχολούμαστε με το φάκελο PNR που είναι δύσκολο για πολλούς ε, γιατί πλέον τα πράγματα δεν ε, είναι πολύ άνετα για μας, αλλά συνεχίζουμε γιατί είναι αρμοδιότητά μας. Αρμοδιότητά μας. Το κύριο στοιχείο είναι η βασική υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, αναλύουμε τα αποτελέσματα των δεδομένων PNR είναι πολύ καλά προσδιορισμένο. Και αν μα ζητήσουν να συμφωνήσουμε με μια οδηγία PNR, το λιγότερο που περιμένουν οι πολίτε είναι αυτέ τι πληροφορίε να ανταλλάσσονται μεταξύ κρατών μελών. Και νομίζω ο κύριο Δεκέχοβε είπε ότι προσπαθούμε να πείσουμε τι μυστικέ υπηρεσίε. Τι εννοείται. Συγγνώμη, σα ακούμε τόσο είναι ώρα. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και έχω και άλλε. Μην αναστατώνεστε. Θα ήθελα να καταλάβω τι εννοείται όταν λέτε να πείσετε τι μυστικέ υπηρεσίε. Είναι δημόσιε αρχέ με κρατική χρηματοδότηση. Αν λέμε σε πολιτικό επίπεδο ότι πρέπει να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών, αυτό θα γίνει. Εντάξει, μερικέ ακόμα παρατηρήσει για την αξιολόγηση τη εργαλειοθήκη. Σε πολλά είπατε και τα χαιρετίζω όμω, γιατί δεν έχει γίνει. Το Κοινοβούλιο ζήτησε αξιολόγηση τη εργαλειοθήκη πριν από τέσσερα χρόνια. Τίποτα δεν έχει γίνει. Και το θεωρώ απαράδεκτο ότι εδώ πέρα μας ε, εξωθείτε να υιοθετούμε νέα μέτρα κάθε φορά και κάθε φορά βλέπουμε ότι τα μέτρα που συμφωνήσαμε την προηγούμενη φορά, με την προηγούμενη επίθεση δεν έχουν υλοποιηθεί. Ήρθε η ώρα αρχίσετε και εσείς να εφαρμόζετε τίποτα. Και το τελευταίο. 50 λεπτά ακούγαμε τους ομιλητές. Είχατε διαμαρτυρηθεί. Εδώ πέρα απλώ χρησιμοποιώ και ασκώ το δικαίωμα του Ευρωβουλευτή. Τίποτα παραπάνω. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ανακοίνωσαν ότι θα ε, περιορίσουν ε, το πρόγραμμα άρση θεωρήσεων. Τι θα ζητήσει σε αντάλλαγμα η Αμερικανική πλευρά, γιατί ξέρω ότι ήδη έχει περάσει μια λίστα επιθυμιών προς ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κυρία Γκίγιομ. Πολλά θέματα αναφέρθηκαν εδώ. Δεν έχω την εντύπωση ότι έκανε και πάρα πολλά το Συμβούλιο. Νομίζω ότι επιταχύνθηκαν τα πράγματα. Ενδεχομένω είναι εντύπωσή μου. Αυτή την αίσθησή μου την ενισχύει το γεγονός ότι οι προτάσεις που διατυπώθηκαν υπάρχουν εδώ και καιρό, έχουν τεθεί επιτάπητος. Δεν έχουμε προχωρήσει πολύ, απλά και μόνο ανακυκλώνουμε το ίδιο πράγμα, ε, το θέμα της, ε, του ξεπλήματος, το θέμα των όπλων κτλ. Νομίζω ότι ε, δεν θα πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας στην αδράνεια του Κοινοβουλίου. Αυτή η ευθύνη καταμερίζεται σε όλα τα, μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων. Ξέρουμε τι έχει γίνει με το PNR. Το καλύτερο παράδειγμα της κοινή αυτής ευθύνη είναι ότι ε, δεν έγιναν και πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Το θέμα, σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, θα επιθυμούσα να αναφερθώ σε δύο προβλήματα. Προσπάθησα να αναφερθώ, στο, να δω τον αριθμό των κατελών που υπάρχει, των ατόμων όλων αυτών που συμβάλλουν σε μία καταγραφή σε μια καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της τρομοκρατίας. Έφτασαν 14. 14 διάφορες ε, καρτέλες. Πραγματικά αναρωτιέμαι αν αυτό αποτελεί ένδειξη αποτελεσματικότητας. Το άλλο θέμα είναι πώς θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε το γεγονός ότι ότι άτομα για τα οποία υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης ε, τον ε, προτέρων ορισμό όλη τους στη ζωή από τότε που πήγαιναν στον υπηαγωγείο αλλά δεν μπορούμε να έχουμε μία ανταλλαγή πληροφοριών. Με άλλα λόγια, πιστεύετε ότι η επεξεργασία των εμπορικών δεδομένων θα υπερισχύσει της ε, επεξεργασίας των δικαστικών και αστυνομικών δεδομένων. Ευχαριστώ κύριε Μπόνη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις ε, παρεμβάσεις σας. Νομίζω ότι απαιτείται μία σαφής αντιτροποκρατική πολιτική στην Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία. Καταρχάς εργαλεία πρόληψης, μέσα πρόληψης, το PNR, το νέο CFTP, ένας ε, καλύτερος ρόλος, πιο αποτελεσματικός ρόλος για την Europol, καθώς και η υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και με αυτόματο τρόπο. Η επεξεργασία των δεδομένων, ο διαρκής έλεγχος της κατάστασης, κατώ βεβαίως από αποδεκτές νομικές ε, βάσεις. Υπάρχουν όμως προβλήματα εφαρμογής αυτών των αρχών. Το πρώτο ερώτημα, αν οι χώρες μέλη πραγματικά είναι έτοιμες να συνεργαστούν στενότερα, να ανταλλάξουν πληροφορίες, να ενδυναμώσουν την Frontex, να εξυγχρονίσουν το σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν. Δεύτερον, σε πολλές χώρες υπάρχει ένα κλίμα προετοιμασίας του δικού τους αντιτροποκρατικού νομικού πλαισίου. Πώς θα μπορούσε να υπάρχει αναρμόνιση αυτών των προσπαθειών. Δεύτερον, ποιο, ποια, ποιος είναι ο πραγματικός συντονιστής, ποιο θεσμικό όργανο αυτών των ενεργειών. Και τέταρτο, δίνουμε τη μάχη μας κατά της τρομοκρατίας, όχι κατά του διαδικτύου. Είναι σημαντικό να βρούμε τα αναγκαία εργαλεία, τους απαραίτητους κανόνες και να βρούμε την ισορροπία μεταξύ αυτών των βασικών θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Η κυρία Ευχαριστώ Πολλά σημεία αναφέρθηκαν από τη συνάδελφό μου, οπότε θα είναι σύντομη η παρέμβασή μου. Σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση εφαρμογή, είχαμε τα έγγραφα για να προετοιμάσουμε αυτή τη συνάντηση. Ο υπεύθυνο είναι Ιντερνετ Καστέρ και αυτό έγινε μετά το Συμβούλιο του Φεβρουαρίου. Δηλαδή, βλέπουμε πόσος χρόνος χρειάζεται για ορισμένα πράγματα. Το έγγραφο αυτό όμως είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ιδιαίτερα το κεφάλαιο 5 που αφορά όλα τα μέτρα που αφορούν τη σωστικοποίηση ε, και την πρόληψη. Αυτό δεν αφορά μόνο την Επιτροπή Λίμπερ αλλά θα πρέπει ε, να μας απασχολήσει θα πρέπει να δούμε αν τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, ανθρώπινο, δυναμικό, οικονομικά μέσα, είναι επαρκή για να επιτελέσουμε το καθήκον μας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε θέματα που έθιξε έφτιαξαν οι συνάδελφοι, δηλαδή το θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ε, διαφόρων υπηρεσιών πληροφοριών. Πέντε χώρες μέλη που έχουν ενεργό συμμετοχή σε ανταλλαγή πληροφοριών ε, είναι πολύ λίγες. Αν σκεφτούμε ότι είμαστε 28 χώρα χώρες μέλη. Όλοι θα πρέπει να έχουμε συμμετοχή. Το άλλο ερώτημα που θα ήθελα να κάνω που αφορά το Συμβούλιο και τις χώρες μέλη θα πρέπει να έχουμε την βεβαιότητα ότι θα γίνουν οι τρεις επόμενες συναντήσεις για το PNR και εύχομαι τα αποτελέσματα της συνάντησης της 20ης Νοεμβρίου να εφαρμοστούν και να αποτελέσουν προτεραιότητα για το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Η Γκόμες. I'm also και εγώ με τη σειρά μου έχω κουραστεί με αυτή τη λειτουργία του PNR, λες και είναι το μαγικό ραβδί. Βεβαίως και εγώ είμαι υπέρ του MNR. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τι διαφορά θα έκανε το PNR. Ε, ήταν γνωστά τα ταξίδια όλων αυτών στην Συρία. Στο Παρίσι δεν πήγαν με αεροπλάνο. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό που χρειαζόμαστε και απευθύνουμε στο Συμβούλιο, χρειαζόμαστε την πολιτική βούληση, την πολιτική ηγεσία και ενώ παράλληλα θα πρέπει να δουλέψουμε με έναν τρόπο ευρωπαϊκό. Ε, ε, συνεχώς επαναρχόμαστε στην εθνική προσέγγιση. Υπάρχουν θέματα για τα οποία δεν ενημερώνονται οι υπηρεσίε πληροφοριών. Θα πρέπει λοιπόν να τα μοιραζόμαστε όλα αυτά. Ακριβώς επειδή λείπει η πολιτική βούληση, επειδή έχουμε αυτές τις εμονές, επειδή υπάρχει θέμα περικοπή περικοπής προϋπολογισμού προσωπικού ε, στον τομέα των υπηρεσιών πληροφοριών, στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών. Για σκεφτείτε το Μόλεμπεκ, το Μόλεμπεκ η ανεργία έχει αγγίξει το 60% και αυτό ε, δεν ε, βοηθάει τα πράγματα βεβαίως. Και βεβαίως για την αντιμετώπιση όλων αυτών χρειάζονται δεξιότητες για να αντιμετωπίζει κανείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να χρησιμοποιεί καλή τη σωστή γλώσσα. Ανεξάρτητα από το τι υπόθηκε μεταξύ την, ε, μετά την επίθεση στο Τσάρλι Εμπρό δεν εφαρμόστηκε. Εμείς έχουμε μία κοινή θέση. Οι χώρες μέλη πάρα πολύ συχνά το έχουν μποϊκοτάρει παρόλο που είναι μια κοινή θέση. Έχουμε ένα πρόγραμμα δράση PRN το οποίο είναι αποδυναμωμένο που δεν εφαρμόστηκε και που οι χώρες ε, μέλη δεν έκαναν τίποτα. Τα όπλα. Τρεις μέρες μετά τις επιθέσεις το Παρίσι δεν ξέρω αν ε, υπάρχει, ε, αν έγινε κάτι σε επίπεδο αστυνομίας και σε επίπεδο όπλων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το θέμα μας δεν είναι η κυνηγή. Νο, έγινε μία αναφορά ότι δεν θα πρέπει να αναμειγνύουμε τους τρομοκράτες με τους μετανάστες. Αυτό κάνουμε. Πώς, τι μπορούμε όμως ε, να κάνουμε δεν υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για να διεξάγονται έλεγχοι. Θα μπορούσαν να, υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες όταν δεν υπάρχουν τρόποι για να ελέγχουμε τους μετανάστες και τους ε, ε τρομοκράτες. Το ξέπλυμα θυμάτων βεβαίως και συμφωνώ ότι θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια έτσι ώστε να εφαρμόζονται τα, όσα έχουμε αποφασίσει. Το, υπάρχει και το θέμα της ε, παρακολούθησης των τραπεζών και αυτό σε σχέση με το ξέπλυμα χρημάτων. Έλεγχη ε, ε, της, Μεταφορά ε, ρευστού. Δεν ξέρουμε, το ξέρουμε ότι οι χρήματα από τι ευρωπαϊκέ τράπεζε περνάνε σε τράπεζε σε όλο τον κόσμο. Τώρα, θα πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο με την Τινησία, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τι συμβαίνει στην ε, Τινησία. Στην Τινησία είχαμε την έκρηξη στο Μουσείο Μπαρντό. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε οποιοδήποτε μέρο. Για πέστε μου όμω με την ε, Τουρκία, η Τουρκία έχει σχέσει με τη Συρία, τη Λιβύη, την Τινησία. Εδώ βλέπουμε ένα διπλό παιχνίδι. Η... Υπάρχουν διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης και οι χώρες μέλη δεν τα αναφέρουν όλα αυτά. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Τουρκία, αλλά αυτό το διπλό παιχνίδι μπορούμε να συνεχίσουμε να το ε, δεχόμαστε. Ο κύριος ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να προσπαθήσω να βάλω λίγο μια αντικειμενική διάσταση στην όλη συζήτηση. Έχω την αίσθηση ότι οι ακραίες καταστάσεις ε, ε, όλο και πιο πολύ συσσωρεύονται. Είτε είναι τρομοκρατικές επιθέσεις, είναι η κρίση των μεταναστών και θα πρέπει να κοιτάξουμε τις αναλύσεις δεδομένων και την ανταλλαγή δεδομένων. Και αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερα είναι κάτι το οποίο ενδεχομένω ε, να είναι σε δευτερεύουσα μοίρα για πολλούς αυτή την εποχή, αλλά είναι το κάτω δικαίου. Θα ήθελα οι σχετικές προδιαγραφέ να πληρούνται για ακραίε καταστάσεις όπου λαμβάνονται ad hoc αποφάσεις. Θα έπρεπε να πω ότι δεν είναι η σωστή στιγμή να σκεφτούμε το τι θα χρειαστούμε στο μέλλον. Χρειαζόμαστε λοιπόν στοιχεία για τη μετακίνηση, για την επικοινωνία, για τις τραπεζικές, ε, για τα τραπεζικά στοιχεία, για να δράσουμε κατά της τρομοκρατίας εδώ στο Κοινοβούλιο, στην ε, σε ό,τι αφορά αυτά τα μέτρα κατά της είναι πριν από λίγες εβδομάδες ήθελε να τα καταργήσει. Θα έπρεπε λοιπόν επί τη αρχής να εξετάσουμε τέτοια ζητήματα και γι' αυτό λοιπόν θα ήταν σημαντικό να γνωρίζουμε. Τι εμποδίζει στην παρούσα φάση την ανταλλαγή δεδομένων. VCC, οι τράπεζες δεδομένων, όλες αυτές. Χρειαζόμαστε τέτοια δεδομένα και για την πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών. Κάτι άλλο που ανέφερα και χθε. Μου απάντησε η συγγήτρια. Αλλά έχω την αίσθηση ότι σε ό,τι αφορά την οδηγία για την προστασία των δεδομένων, την οποία επεξεργαζόμαστε στην παρούσα φάση και λέμε ότι τα κράτη-μέλη δεν μας έχουν ε, διαβιβάσει δυσκολίες, νομίζω ότι κανείς δεν έχει κάτσει να κοιτάξει κατά πόσον όλα αυτά τα οποία συμφωνούμε στο πλαίσιο του, της νομοθεσίας αυτής ε, έχουν εφαρμογή σε μια ακραία κατάσταση σε ένα κράτος δικαίου. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τι δεδομένα χρειαζόμαστε στην τελική ανάλυση. και κατά πόσον δημιουργούνται νομικά μέσα τα οποία καλύπτουν και τέτοιε ακραίε καταστάσει. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο, Να δώσω το λόγο στους συναδέλφους μάλλον και να σας καλέσω εκ νέου να τηρήσετε το όριο των δύο λεπτών. Εγώ φταίω, αλλά έχουμε καθυστερήσει. Κυρία Λόρεσταν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τους ε, τρεις ομιλητές και να τονίσω ότι σε αυτή την κατάσταση μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις όλοι θεωρούμε ότι έχει αλλάξει το πλαίσιο εργασιών μας. Και πρέπει να εξετάσουμε και να αναλογιστούμε όλη την κατάσταση, όλο το πλαίσιο. Αυτό που δεν άκουσα στις ε, παρουσιάσεις είναι κάτι το οποίο Έφτιαξε ο κύριο Βόσα, βεβαίω με την αρνητική σκοπιά, το θέμα τη προστασία δεδομένων. Γιατί ο κύριο Δεκέρκοβε μίλησε για πολλά δεδομένα, βάση δεδομένων, όλα αυτά με τα δεκαλικά αποτυπώματα κτλ. Αλλά ούτε λέξη για την προστασία δεδομένων. Μπορεί κάποιο να έχει τη δυνατότητα ότι στην νέα αυτή κατάσταση η προστασία δεδομένων πλέον δεν έχει καμία σημασία. Πολλοί έτσι σκέφτονται. Πρώτα η ασφάλεια και μετά τα ανθρώπινα δικαιώματα και προστασία δεδομένων είναι κάτι το παροχημένο. Εγώ θεωρώ ότι είναι το αντίθετο που ισχύει. Σε αυτήν την κατάσταση οι βασικές αρχές, αξίες και ελευθερίες είναι αναπόσπαστο τμήμα του κράτους δικαίου, κύριε Βος. Και γι' αυτό πρέπει πραγματικά να τα εξετάσουμε όλα αυτά και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο γιατί ακριβώς αυτό τόνισε ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο πλαίσιο το στομότερο δυνατόν. βλέπουμε και από τις ομιλίες σας αλλά και γενικά ότι υπάρχει αυτό το παράδοξο μεταξύ της κοινοτικής μεθόδου και θέλουμε και αυτές τις κοινέ πολιτικές αλλά και συνθήκη ε, όλα αυτά τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και δημόσιας ασφάλειας εναπόκειται στα κράτη-μέλη. Εντάξει, δεν χρειάζεται να γίνει και αιμονή το ότι έχουν διαφορετικέ θεωρίε στα κρατημέλη. Ισχύει αυτό σε έναν βαθμό. Το Βέλγιο βλέπουμε ότι έχει διαφορετική ερμηνεία τη ασφάλεια και θεώρηση τη ασφάλεια από ότι η Γαλλία, για παράδειγμα, παρότι είναι γειτονικέ χώρε. Πόσο μάλλον ε, χώρε ε, στα ανατολικά σύνορα σε σχέση με χώρε ε, στα νότια σύνορα. Πρέπει όμω να βρούμε μια κοινή θεώρηση της Ευρωπαϊκή δημόσια ασφάλεια για να έχουμε μια αποτελεσματική κοινή πολιτική. Γιατί τώρα, για παράδειγμα, συζητούμε μία οδηγία, αλλά πρέπει να δούμε τι ακριβώς εννοούμε με μια κοινή ευρωπαϊκή δημόσια ασφάλεια. Και το δεύτερο που θα ήθελα να τονίσω. Ναι, είπατε ότι πρέπει να υπάρχει πρόληψη και χρειαζόμαστε την παιδεία γι' αυτό. Πρέπει να κατανοήσουμε τι είδου ε, βασικές αξιο... Ε, δεξιότητες χρειάζονται. Και εγώ είμαι καθηγήτρια επικοινωνία. και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, βαθύ, διαπολιτισμικό και διάθρησκευτικό πρόβλημα. Το νέο αφήγημα δεν είναι μόνο ένα μότο Χρειαζόμαστε ειδικού εμπειρογνώμονε, ειδικού στην ιστορία, στη θρησκεία και το Ναι, η επιστήμη τη πληροφορία καλή είναι, καλέ και αστυνομικέ αρχέ. Αλλά αν δεν γνωρίζουμε σε βάθο του ε, λόγου του οποίου συμπεριφέρεται κανεί έτσι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Κοινωνικέ επιστήμε και οι ανθρωπιστικέ επιστήμε γενικά πλέον θεωρούνται κάτι το περιττό και το άχρηστο και πάντα μιλούμε για τις ε, θετικές επιστήμες και την τεχνολογία. Αλλά τώρα πρέπει να καταλάβουμε ότι και οι ανθρωπιστικές επιστήμες θα πρέπει να μας απασχολήσουν περισσότερο για να λύσουμε ακριβώς αυτά τα ε, πολύ σοβαρά ζητήματα. Συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος, όλοι οι ομιλητές υπερβαίνουν ε, το χρονικό τους όριο. Βεβαίω αυτό είναι αναπόφευκτο γιατί υπάρχει μία σωρία πολύ σημαντικών ζητημάτων που εξετάζουμε εδώ. Γι' αυτό ήθελα και να δώσω το χρόνο στους συναδέλφους να τα αναφέρουν όλα τους τα ερωτήματα. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στους ε, ομιλητές. Θα τροποποιήσουμε την εμείς διάταξη για να έχετε περισσότερο χρόνο. Συνάδελφοι, λίγη πειθαρχία, αν μπορείτε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. μεγάλη χαρά βλέπω ότι συμφωνούμε πόσο επίγον είναι να έχουμε το PNR. κάλιο αργά παρά ποτέ, όπως λένε. και βλέπω ότι ε, και με ενδιαφέρον βλέπω ότι κάποιοι παίρνουν το λόγο και λένε τα αντίθετα αυτά που έλεγα πριν μερικά χρόνια. Μπορείτε να δείτε και τα πρακτικά. Τώρα, τι θα γίνει με το PFTP αν πραγματικά ε, έχει παρεμποδιστεί η διαδικασία και αν τελικά θα καταλήξουμε σαν ευρωπαϊκό PFTP. Και το ερώτημα των ε, χορηγιών και δωρεών που έρχονται από συγκεκριμένα κράτη ε, και μεταφιέζονται ως φιλανθρωπίες. Πολλές φορές έρχονται και από πολλές αραβικές τράπεζες. Όπως είπε και η κυρία Γκόμες, σίγουρα υπάρχει και χρηματοδότηση τρομοκρατική. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μας απασχολήσει η ριζοσπαστικοποίηση και η παιδεία είναι κρίσιμη σημασίας είναι μια έκτακτη ανάγκη αυτό που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Μια επίγουσα κατάσταση. Η κοινή πολιτική άμυνας και, και εδώ είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Δεν υπάρχει πολιτική δέσμευση για να υπάρξει αυτή η πολιτική. Όμως το πλέον σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι οι πολίτε μας να καθησυχαστούν. Χώρε όπω η Ισπανία που έχει υποφέρει πολύ από την ε, τρομοκρατία ίσω είναι καλύτερα προετοιμασμένη από ότι σε άλλα κράτη-μέλη που το επίπεδο ετοιμότητα δεν είναι ε, αρκετά υψηλό. Κύριε Ντεγκαρχόβε, πρέπει να εργαστούμε περισσότερο και να δώσουμε περισσότερα χρήματα στι αστυνομικέ αρχέ. θα πρέπει οι αστυνομικέ αρχέ, οι δικαστικέ αρχέ και ούτω καθεξή να είναι σωστά προετοιμασμένε για αυτή τη νέα απειλή που έρχεται από παντού. Δεν υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών αυτή τη στιγμή και ε, διστάζουμε κιόλα να προβούμε σε αυτήν την ανταλλαγή πληροφοριών. Κάποιε φορέ υπάρχει και δυνατότητα ε, ικανότητα ή ετοιμότητα μάλλον. Δεν κατακρίνω τι ικανότητέ του, αλλά εδώ πέρα δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά είναι αυτή η νέα βαρβαρότητα Τη τρομοκρατίας. Ευχαριστώ ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγγνώμη, καθυστέρησα. Ίσως επαναλάβω πράγματα που έχουν ήδη υποθεί. Όλα τα ερωτήματά μου αφορούν την αναγκαιότητα ενίσχυση τη ανταλλαγή πληροφοριών. Πρώτον, στη χώρα μου, αλλά και στο Κοινοβούλιο εδώ, πολλές φωνές ζητούν την εισαγωγή ενός ε, μιας υπηρεσίας πληροφοριών, κάτι αντίστοιχο με μια CIA. Ποια είναι η θέση σας ε, ως προς αυτό. Θεωρείτε ότι πρέπει να έχουμε νέο θεσμικό όργανο, να μεταμορφώσουμε και να αλλάξουμε την Europol. Ε, τι θα γίνει. Δεύτερον, μίλησατε για νομοθετική πρόταση που θα υποβληθεί σύντομα για την διασταύρωση ε, βάσαν δεδομένων με την Europol και για το SIS2. Ε, όμως ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, πότε θα γίνει αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Τρίτον, για το PNR. Διάβασα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, μιλούν για ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό PNR. Εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό PNR. Είναι εθνικά PNR τα οποία οργανώνονται με το ίδιο μοντέλο αλλά να αναφέρω το εξή. Έστω ότι υπάρχει ένας τρομοκράτης που φεύγει με το τρένο από το Παρίσι, ε, έρχεται Βρυξέλλες, παίρνει το αεροπλάνο, πάει ε, στην Τουρκία. Με το εθνικό PNR οι Βέλγοι είναι αυτοί που καταχωρίζουν τα δεδομένα. Όμως αν δεν έχει μπει στο ΣΥΣ, ε, αν δεν υπάρχει δηλαδή συστηματική πληροφόρηση για να ξέρουμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, τότε τι νόημα έχει. δεν πρέπει να υπάρχει υποχρέωση για όλα τα κρατημέλη να βάζουν αυτά τα δεδομένα στο ΣΥΣ και στη βάση δεδομένων της Europol. Να βάζουν αντί αυτά τα πρόσωπα που είναι ύποπτα για τρομοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητήσαμε εκτενώς το θέμα των μέτρων ασφαλείας και του PNR κτλ. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα γιατί θα πρέπει να δίνουμε στους ανθρώπους ένα αίσθημα ασφαλείας. Πιστεύω όμως ότι συζητάμε πολύ λιγότερο για θέματα ολοκλήρωσης και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ομάδες εργασίας, αλλά χρειαζόμαστε και αυτά θέματα εδώ. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα σημείο τι γίνεται σε ό,τι αφορά την διασύνδεση μεταξύ ανεργίας, περιθωριοποίησης κοινωνικής και της αίσθηση απομόνωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο θέμα εκπαίδευσης, παιδείας. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα. Υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα. Κύριε Τεκέρχοφ, αναφερθήκατε στη σχέση μεταξύ ε, μετανάστευσης και τρομοκρατίας και είπε ότι είναι ένας τοξικός συσχετισμός. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που το χρησιμοποιούν αυτό και συνεπώς θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα ποιο είναι το πρόγραμμα της Επιτροπής ε, τι έχει σκοπό να κάνει η Προεδρία για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και κάτι ακόμα. Υπάρχουν μέλη σε αυτό το κοινοβούλιο που χρησιμοποιούν την ίδια τοξική ε, συλλογιστική. Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε αποτελεσματικές πολιτικές ε, όταν υπάρχουν μέλη που συνεχίζουν να κάνουν αυτή την τοξική διασύνδεση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επικεντρώσω την προσοχή μου σε δύο σημεία επειδή ο χρόνος πιέζει. Το πρώτο που δεν αναφέρθηκε είναι ο δικαστικός κλάδος. Για παράδειγμα στην Ιταλία συνελήφθησαν άτομα ύποπτα για τρομοκρατικές ε, πράξεις είτε διότι αντάλλαξαν ε, πληροφορίες στο ίντερνετ ή για κάτι άλλο αλλά που αποφυλακίστηκαν αμέσως. Θα ήθελα να γνωρίζω σε ό,τι αφορά το δικαστικό σώμα υπάρχει κάποια συνειδητοποίηση του πώς έχουν τα πράγματα πριν το Παρίσι και μετά το Παρίσι. Ένα άλλο θέμα, μιλάμε για intelligence, για ανταλλαγή πληροφοριών. Οι δρομοκράτες ήταν στις Βρυξέλλες, δεν ήταν σε απίθανα μέρη σε περιοχές που δεν μπήκαν ποτέ οι δυνάμεις διωξη με εξαίρεση τις τελευταίες επιδρομές της αστυνομίας. Κάτι τελευταίο, η μουσουλμανική κοινότητα εδώ δεν μιλάμε για θρησκεία όταν έχουμε να κάνουμε με την τρομοκρατία. Δεν υπάρχει θρησκεία. Οι τρομοκράτες είναι κάτι άλλο. Και η σημασία του διαλόγου με τη μουσουλμανική κοινότητα είναι ότι δεν χρησιμεύει ε, το να ελέγχουμε τις μαζικές εκδηλώσεις χρησιμεύει να υπάρχει έλεγχος επί των χωρών μελών, επί των κέντρων που γίνονται κηρύγματα σε μία χώρα που δεν είναι μια γλώσσα κοινωνική, κοινοτική σημεία που δεν υπάρχει θρησκεία, υπάρχει κάτι άλλο. Από τις μουσουλμανικές κοινότητες ε, δεν ε, ε, ζητάμε μία ανάληψη δέσμευσης. Θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη επαγρύπνηση σε ό,τι αφορά τους νέους. Εκείνοι ξέρουν πολύ καλύτερα από μας τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινότητα που ζουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απευθύνω το ερώτημά μου στον Τύριο Κιγόλα. Γιατί εσείς είστε ο συντονιστής για θέματα τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαίνει ότι δεν είστε επίτροπο για κοινωνικά θέματα. Ένα θέμα που είναι σημαντικό όταν καλούμεθα να καταλάβουμε τι πήγε καλά, ε, άσχημα, πού οφείλεται αυτή η τροτότητα σε αυτή την ε, απειλή που προσλαμβάνει τη μορφή του φανατισμού και εξισλαμισμού. Εσείς είστε ο συντονιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα τρομοκρατίας και αν κάτι είναι, μάθαμε σαφώς μετά από τις τρομερές εμπειρίες είναι ότι υπήρξε έλλειψη συντονισμού. Όταν όμως διαβάζουμε τις ειδήσει, όταν κοιτάμε τα νέα στην τηλεόραση ε, που αφορούν το τελευταίο Συμβούλιο, αυτό που βλέπετε είναι να επικρίνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κατάφερε να ε, υιοθετήσει τους κανόνες για το PNR, το μπλοκάρισε. Δεν είναι αλήθεια όμως αυτό. Υπάρχει κάποια αυτοκριτική μέσα στο Συμβούλιο όταν τίθεται το θέμα της έλλειψης συντονισμού ή γίνεται κάποια αυτοκριτική στο Συμβούλιο όταν τίθεται το θέμα της έλλειψη πληροφοριών, έλλειψης ε, ανταλλαγής πληροφοριών σε ό,τι αφορά θέματα ασφαρία, σε ό,τι αφορά ε, υπηρεσίες πληροφοριών. Υπάρχει κάποια στρατηγική για τη δημιουργία ενός μιας καινούρια μονάδας πληροφοριών ε, ή τουλάχιστον και κάτι, κάτι βασικό για να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να ε, δυναμώσουμε, να ε, μπορέσουμε να, να τα προλάβουμε όλα αυτά σκέφτεστε κατά κάποιο τρόπο να επενδύσετε στη μονάδα πληροφοριών που υπάρχει τώρα και για την οποία είναι υπεύθυνη η εξωτερική πολιτική. Έχετε κάποια σκέψη να τα επεξεργαστείτε όλα αυτά. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Δύσκολη ερώτηση που κάνατε. Δύο μιλήτες. Ο κύριος Δέτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εν συντομία να πω χάρηκα για όσα άκουσα. Σε επίπεδο κοινοβουλίου, σε ό,τι αφορά αυτή την κολλησιεργία στην οποία έγινε αναφορά, θα ήθελα να κάνω μια έκκληση. Να απευθύνω μια έκκληση έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουμε ότι εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο κατοίκον σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, κάτι που έχει άμεση σχέση με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ θα ήθελα να στηρίξω τον αγώνα που δίνεται και σε ό,τι αφορά τους κώδικες αποκωδικοποίησης και σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο. Πριν να επιβεβαιωθεί κανείς ένα αεροπλάνο, θα μπορούσατε να μας πείτε τι θα μπορούσε να κάνει κανείς κάτι το απτό. Τι θέλετε να γίνετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Το πρόβλημα καταρχάς είναι η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που επήγει. Χρειάζεται χρόνος για την εφαρμογή των μέτρων. Αν σταματήσει σύντομα η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, θα μπορέσουμε να βάλουμε τέλος τα όσα συμβαίνουν. Η ε, νομιμοποίηση παράνομων προσόδων είναι ένα θέμα σε πολλές χώρες. Η δίμευση είναι ένα άλλο θέμα. Ε, η δίωξη ε, όλων αυτών θα πρέπει να γνωρίζουμε όλες τις συναλλαγές ε, που λαμβάνουν χώρα. Οι συναλλαγές θα πρέπει να γίνονται μέσω τράπεζας. Οι υπηρεσίε πληροφοριών θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και μερικές από αυτές συνεργάζονται. Όχι όλες βέβαια, γιατί οι μερικές ε, δεν εμπιστεύονται τις άλλες. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει το Συμβούλιο ή οι χώρες μέλη. Γιατί αν η μία υπηρεσία πληροφοριών δεν εμπιστεύεται την άλλη, δεν ξέρω τι μπορείτε να κάνετε. Μπορεί να γίνει κάτι στο Συμβούλιο. Το τελευταίο σημείο αφορά το θέμα των ε, θεωρήσεων. Ξέρω ότι υπεγράφει μία συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για ένα ελεύθερο καθεστώς θεωρήσεων. Το Κοινοβούλιο δεν έδωσε ακόμα τη σύμφωνη γνώμη του συζήτησα το θέμα με τον πρόσωπο, αντιπρόσωπο της μόνιμης αντιπροσωπείας βεβαίως ε, ε, επικοινώνησε με την Λύπε, το ρώτημά μου ήταν δεχτήκατε πρόσφυγες είπε όχι γιατί του είπα ε, εγκρίνεται αυτό το καθεστώς σε χώρες που είναι ασφαλείς και που θα μπορούσαν να δεχτούν πρόσφυγες και να ασχοληθούν με αυτούς Νομίζω ότι θα πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη όταν τεθεί το θέμα ενώπιον της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Επέτρεψα και στους συναδέλφους που έφτασαν καθυστερημένοι να κάνουν ορισμένα σχόλια. Ήθελα μόνο να ξεκαθαρίσω, επειδή ακριβώς είναι τόσο περίπλοκη η συζήτηση, επέτρεψα στους συναδέλφους να μιλήσουν όσο ήθελαν χωρίς να τους διακόψω. Και θα τροποποιήσω ένα λόγο στην διάταξη, γιατί είναι τόσο σημαντική και επίκαιρη αυτή η συζήτηση και σχεδόν όλοι όσοι ήρθαν σήμερα στη συνεδρίαση πήραν τον λόγο. Ήθελα μόνο να σχολιάσω αυτό που είπε ο κύριο Λόπεθ Αγγιλάρ. Αρκετά μέλη αναφέρθηκαν και συνάδελφοι θα έχετε πολύ χρόνο να απαντήσετε, δεν θα σας περιορίσω καθόλου στο χρόνο. Επομένω, αυτή την διαφοροποίηση ε, ανάμεσα σε αυτά που κάνει ε, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, το Συμβούλιο και πώς ε, όλα αυτά γίνονται αντιληπτά. Δεν είναι κάτι καινούργιο όμως αυτό. Η απόφαση Προύμ και το 2005. Εφτά κράτη-μέλη ούτε καν μπαίνουν στον κόπο ε, να ανταλλάξουν δεδομένα DNA. Άλλα οχτώ ε, δεν ανταλλάζουν τελικά αποτυπώματα. Τώρα μιλούμε για μια νέα νομοθεσία για τα πυροβόλα όπλα και μας, ζητού... μας έχετε ζητήσει να το υιοθετήσουμε. Εμείς τη δουλειά μας την κάνουμε ό,τι και αν γίνει, εμείς σκληρά θα εργαστούμε. Μην νομίζετε λοιπόν ότι εμεί δεν είμαστε εταίροι και δεν συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο για την καταπολέμηση τη Δημοκρατία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα ήθελα και εγώ να το αναφέρω ω Πρόεδρο. Όμω. Τα μέλη ήθελαν να, να μας ξεκαθαρίσετε ακριβώς τι κάνει το Συμβούλιο από πλευρά επιβολή. Από το 2014 είχατε δυνατότητα να υλοποιήσετε την απόφαση Πλουμ. Και αυτό θα πρέπει να το ξέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήθελα λοιπόν να κάνω αυτά τα σχόλια και να σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε όσο θέλετε. Και θα τροποποιήσουμε για την ίδια διάταξη. Παρακαλώ από πλευρά ε, Λουξεμβουργιανής Προεδρίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλους ε, τους ευρωβουλευτές ε, για τις ε, ερωτήσεις και παρατηρήσεις τους. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να απαντήσω σε αυτό που μόλις είπατε. Νομίζω ότι το Συμβούλιο και πιο συγκεκριμένα η Λουξεμβουργική Προεδρία θεωρεί πραγματικά το Κοινοβούλιο πολύ σημαντικό εταίρο πάρα πολύ σημαντικό εταίρο σε, όλα όσα υλοποιούμε. Πράγματι, η ευθύνη για την εφαρμογή αφορά τα κράτη-μέλη και τις υπηρεσίες τους. Όμως εδώ πέρα όλοι μαζί εργαζόμαστε από κοινού. Όλοι οι φορείς σε όλα τα επίπεδα. Εμείς έχουμε φτάσει στο τέλος της προεδρίας μας, στο τέλος της θητείας μας. Δεν έχει έρθει βέβαια η ώρα ακόμα του απολογισμού, αλλά μπορώ να σας πω ότι θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε με το Κοινοβούλιο όπως εξαιρετική ήταν συνεργασία μας στους τελευταίους μήνες και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα συνεχιστεί και στους μεγάλους φακέλους που έχουμε ενώπιόν μας όπως είναι το PNR, προστασία δεδομένων για να φέρω μόνο δύο τομείς. Ένα πρώτο στοιχείο σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες. Με δύο λόγια μόνο. Δεν θέλω να θεωρήσω ότι πρόκειται για δικαιολογία. Είναι μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που μας έχει επιβληθεί από τη συνθήκη. Αυτό που αποκαλούμε εθνική ασφάλεια, με αυτόν τον όρο καλύπτεται ε, στη συνθήκη το intelligence, είναι εκτός αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, αν εξετάζουμε ζητήματα μυστικών πληροφοριών ε, στο Συμβούλιο, όχι. Γιατί η συνθήκη μας το απαγορεύει να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Είναι τομέας που δεν εμπίπτει στο δικό μας πεδίο αρμοδιοτήτων. Αυτό βεβαίως δεν απαγορεύει στις ε, εθνικές υπηρεσίες να συνεργαστούν μεταξύ τους. Και είμαι πεπισμένος ότι και ο Ζήλ θα πει κάτι παραπάνω για αυτό το ζήτημα γιατί μέσω και των δικών του προσπαθειών έχουμε τη σύνδεση μεταξύ των όσων συμβαίνουν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσων συμβαίνουν εκτός. Υπάρχει μια σημαντική πτυχή της πάλι κατά της τρομοκρατίας που συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το κοινοτικό δίκαιο. Πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Άκουσα πολλά σημεία κριτικής. Ε, Είπατε ότι τα κράτη-μέλη δεν κάνουν τίποτα, δεν ανταλλάζουν πληροφορίες, δεν χρησιμοποιούν τις βάσεις δεδομένων. Νομίζω ότι έτσι τα προσφέρεστε λίγο υπεραπλουστευμένα τα πράγματα. Έχουμε το σύστημα SIS ε, της ΕΝΚΕΝ που είναι πραγματικά πετυχημένο ε, γιατί και τροφοδοτείται και χρησιμοποιείται. Έχουμε και άλλες βάσεις δεδομένων, όπως είναι βάση δεδομένων Interpol για τα ε, κλεμμένα διαβατήρια. Ναι, πράγματι δεν αξιοποιούνται επαρκώς. Θα αναγνωρίζουν και τα κράτη-μέλη αυτό. Αυτό ισχύει. Κάνουμε κριτική και αυτοκριτική και στο Συμβούλιο και οι Υπουργοί μετά το Συμβούλιο Τζάι ανέφεραν ότι αναγνωρίζουν πως πρέπει να αναλάβουμε δράση. Και πράγματι αν και τα συμπεράσματα, η έμφαση δίνεται όχι στα νέα μέτρα, αλλά στην υλοποίηση των υφιστάμενων μέτρων. η βάση δεδομένων όπως αυτή είναι της Interpol ε, χρησιμοποιείται εκατοντάδες ε, χιλιάδες φορές από τα κράτη-μέλη. Πράγματι, βεβαίως, ε, υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Το ίδιο ισχύει και για την απόφαση πριν. Είναι ένα σύστημα το οποίο υλοποιείται πολύ αργά, αυτό είναι αλήθεια, όχι αρκετά γρήγορα, αλλά είναι περίπλοκο το σύστημα γιατί καλύπτει όχι μόνο τις εθνικές βάσεις δεδομένων, 28 εθνικές βάσεις δεδομένων, αλλά και διαφοροποιημένες βάσεις δεδομένων σε τομείς ιδιαίτερα ευαίσθητους, όπως είναι τα δεδομένα DNA ή δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τώρα, για να κάνουμε αυτή τη διασύνδεση μεταξύ κρατών μελών, αλλά να κάνουμε και του ελέγχου για την τήρηση των προτύπων προστασία δεδομένων, όλα αυτά είναι σύνθετο εγχείρημα. Παίρνουν χρόνο, παίρνουν πόρου, οικονομικού και ανθρώπινου. για το PNR. Πολύ αναφέρθηκα σε αυτό πράγματι. Και οι υπουργοί έθιξαν αυτό το ζήτημα και όχι μόνο μετά τις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά και πριν. Πράγματι, τα τρία στοιχεία που εμπεριέχονται στα συμπεράσματα είναι τα κύρια στοιχεία για το Συμβούλιο σε τη φορά της διαπραγματεύσεις. Ταυτόχρονα όμως οι Υπουργοί υπογράμμισαν την βούλησή τους στην ίδια προθεσμία να ολοκληρωθεί και μεταρρύθμιση για την προστασία δεδομένων. Το επεσήμανα και χθε. Σε ό,τι αφορά την οδηγία για την προστασία δεδομένων, μία παρατήρηση μόνο από πλευρά Συμβουλίου Κρατών Μελών αυτή η ισορροπία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διαπραγμάτευση είναι μια καλή ισορροπία για να διασφαλίσουμε την προστασία δεδομένων και να διευκολύνουμε και τη, τη δουλειά των αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Για την ιστορία να σας πω ότι ε, στην αντιπροσωπεία μας έχουμε και την διευθύντρια των αστυνομικών αρχών μαζί μας, ακριβώς για να διασφαλίσουμε ότι και η αστυνομία θα αξιοποιήσει αυτά τα συστήματα και δεν θα παρεμποδίσουμε ε, το έργο της. Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων τώρα. Ήθελα να θίξω δύο σημεία. Πρώτον, εάν υπάρχει αλληλοβοήθεια μεταξύ κρατών μελών για την αντιμετώπιση δυσκολιών. Ναι. Για παράδειγμα, έλλειψη μηχανημάτων Eurodac στην Ελλάδα, στα νησιά, γιατί βεβαίω είναι και τεράστιες ερωές. Υπήρξε μια πρωτοβουλία της Προεδρίας που συνεργάζεται με τα κρατημέλη για να αντιμετωπίσουμε αυτή την έλλειψη έχει γίνει αυτό εν μέρη και εξακολουθούμε να το εξετάζουμε. Δεύτερον, για τους Ευρωπαίους πολίτες. Γιατί το, το Συμβούλιο θεωρεί ότι χρειάζεται ε, συγκεκριμένη αναθεώρηση ε, στη Σέγγεν. Γιατί αυτή τη στιγμή ε, οι πολίτες που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα της Σέγγεν ελέγχονται σε ελάχιστο βαθμό. Ε, δηλαδή ελέγχουμε το διαβατήριό του, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε συστηματικό έλεγχο στη βάση δεδομένων αν αυτό το διαβατήριο είναι πλαστό ή κλεμμένο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε συστηματικά αν πρόκειται για καταζητούμενο. και εκτιμένο. αυτό απαγορεύεται ρητός. Λέμε ότι γίνεται μη συστηματικός έλεγχος. Αυτό είναι το διακύβευμα ουσιαστικά. Κατανοώ ότι υπάρχουν, ε, μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, αλλά ήθελα μόνο να το διευκρινίσω. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε συστηματικούς ελέγχους για το κατά πόσο αυτό το πρόσωπο βρίσκεται στο SIS, ε, εάν κρεμεί ένταλμα σύλληψής του, αν είναι πιθανός ε, τρομοκράτης. Για το πρόγραμμα άρσης θεωρήσεων και τα αιτήματα των Αμερικανών ως Προεδρία δεν έχουμε λάβει γνώση ενός συγκεκριμένου ε, καταλόγου επιπλέον απαιτήσεων από πλευράς Αμερικής. Για το ΣΕΜΠΕΡΕΝ είναι ένα στοιχείο το οποίο εξετάζουν τα κράτη-μέλη, ιδίως ό,τι αφορά τις εξωτικές ε, ουσίες. Γίνονται, γίνεται τεράστια δουλειά και για και στο ιστορικό επίπεδο και στο Λουξεμβούργο ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει πολύ, έχουμε επενδύσει πολλά γιατί έχουμε και σημαντική μεταφορά εμπορικών πόρων μέσω εναέριων οδών. Κάτι τελευταίο για την πρόληψη. Εκτός και αν κάνω λάθος, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά τώρα τον, στις 20 Νοεμβρίου που οι Υπουργοί ασχολήθηκαν ενδελεχώς με το ζήτημα της ε, πρόληψης της ρίζοσπαστικοποίησης. Νομίζω ότι μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε μια πολύ σημαντική δουλειά και με αυτή τη συνδιάσκεψη που έγινε που επέτρεψε να συγκεντρωθούν οι Υπουργοί Δικαιοσύνης αλλά και πολλοί ειδικοί σε αυτόν τον τομέα. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο ο τομέας και σε τοπικό, σε περιφερειακό επίπεδο όπου γίνεται πολύ σημαντική δουλειά από τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Νομίζω ότι είναι ένα μακρόπνοο σχέδιο ε, και οι Υπουργοί αναγνωρίζουν τη σημασία του, είναι διατεθειμένοι να το στηρίξουν και από πλευράς οικονομικών πόρων, κατάρτισης, δικτύωσης ε, των ε, φορέων για να υπάρχει μια καλή ανταλλαγή εμπειριών γιατί υπάρχει σημαντική πείρα σε ορισμένα κράτη-μέλη και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής αυτών των εμπειριών για να αποφεληθούν όλοι και να έχουν την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Μεταξύ άλλων και στον τομέα της παιδείας ε, ως τελευταία παρατήρηση. Σας ευχαριστώ και για το θέμα που θίξατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την Προεδρία για την ε, προσπάθεια που καταβάλουν και στους τρεμερεί διαλόγους. Ο κ. Τικερκόπ ε, έχει το λόγο. Τζίλ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα επικεντρωθώ στι απαντήσεις μου σε δύο βασικά ζητήματα. Γιατί πολλέ και εξαιρετικέ ήταν οι ερωτήσει που ακούσαμε, λυπάμαι να δεν απαντήσω σε όλες. Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο είναι ο καλύτερος τρόπος να τα απαντήσω. Καταρχάς, ε, ε, για την ανταλλαγή πληροφοριών και κατά δεύτερον για την πρόληψη. Να επαναλάβω για την ανταλλαγή πληροφοριών αυτά που είπε ο συνάδελφο. Είτε μα αρέσει είτε όχι, οι συνθήκε έχουν όπω έχουν. Αυτά είναι απόφαση των κρατών μελών. Η εθνική ασφάλεια αποτελεί αρμοδιότητα αποκλειστική των κρατών μελών ακόμα. Προσπαθώ να οικοδομήσω γέφυρε μεταξύ αυτή τη κοινότητα που λειτουργεί εκτό τη Ένωση και των μηχανισμών και εργαλείων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι απλό όμω. Και δεν είναι τυχαίο τότε στη συζήτηση για τη συνθήκη της Λισαβόνας κάποια κράτη-μέλη επέμειναν να μείνουν αυτά εκτός του πλαισίου της Ένωσης. Αλλά αν η εθνική ασφάλεια θα πρέπει να ρωτηθούμε κατά πόσο θα πρέπει σε κάποια φάση να δημορφωθεί στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής ασφάλειας. Είναι παγκόσμιες οι προκλήσεις πλέον. Και όσο πιο πολύ αναπτύξουμε την, το κύρος ε, και την εμπιστοσύνη που έχει ο κόσμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο πιο πολύ θα είμαστε σε θέση να δώσουμε κίνητρα ε, στο κρατημέλη να ενταχθούν στην ευρωπαϊκό πλαίσιο. Κατά δεύτερον, αναφέρθηκα σε αυτή τη θεσμική σχιζοφρενία, αλλά η συνθήκη της Λισαβόνας είναι αρκετά πρόσφατη κατά κάποιο τρόπο. 15 χρόνια νομίζω ε, εργάζομαι για να οικοδομήσουμε τον ε, τρίτο πυλώνα, ελπίζοντας ότι θα μετακινηθεί στον πρώτο πυλώνα. Τώρα λοιπόν έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει τις διαδικασίες επί παραβάσης, θα ασκήσει νομική πίεση στα κρατημέλη. Το 2005 διαπραγματευτήκαμε τις σχετικές συμφωνίες και επιβλήθηκε ε, νομική υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να ενημερώνουν τη Γύρω και τη τζαστ για οποιαδήποτε τέτοια εκκρεμή ποινική υπόθεση και δίωξη. Και θα πρέπει να αναγνωρίσω ότι με εντυπωσιάζει η ηγεσία που επιδεικνύει η Επιτροπή Juncker γιατί θέλουν πραγματικά να ηγηθούν στη διαδικασία αυτή και πολλές εξαιρετικές προτάσεις υποβάλλουν. Θα έχουμε για τη φυλακή, σύντομα μια τέτοια πρόταση. στη Γενική Διεύθυνση Home. Πρακτικά τι γίνεται. Προστατεύουμε ήπιους στόχους και χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία και τις μυστικές υπηρεσίες. Είναι πάρα πολύ ασαφής ε, η διαδικασία αυτή. Προσπαθούμε λοιπόν να βάλουμε όλους τους ε, ανθρώπους ε, που εμπλέκονται σε αυτό σε διάφορα τομείς. Για παράδειγμα, την αεροπορία. Αυτό το έθεσε και ο Ολιβιέ. Προσπαθούμε λοιπόν να οικειοποιηθούμε αυτές τις κοινότητες. Αυτά δεν πρόκειται να αλλάξουν σε μία νύχτα ασφαλώς. Και αυτό με οδηγεί στο τρίτο μου ζήτημα, ότι υπάρχει πληροφορία αν υπάρχει εμπιστοσύνη. Και δεν υπάρχει ενδεχομένως επαρκής εμπιστοσύνη μεταξύ των 28. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να εργαστούμε και νομίζω 30 χρόνια πήρε από τον στον Edgar Hoover να περάσει το FBI σε ένα ομοσπονδιακό κράτος. Εμείς δεν είμαστε καν ομοσπονδιακό κράτος. Καταλαβαίνετε τη δυσκολία. Γιατί δεν χρησιμοποιούνται πιο πολλά στοιχεία στο 36.3 του ΣΥΣ ε, για τους ε, τζιχαντιστές. Κοιτάξτε, η διαδικασία είναι πάρα πολύ δύσκολη και οι μυστικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ασφαλείας χρησιμοποιούν τις μεθόδους τους και συλλέγουν ε, κομμάτι-κομμάτι τις πληροφορίες. Έχουν κάποια στοιχεία. Αυτό δεν ε, σημαίνει ότι ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει στην Συρία. Ξέρουμε ότι υπάρχει ριζοσπαστικοποίηση σταδιακή, ότι υπάρχει πιθανότητα ταξιδιού κτλ. Προσπαθούμε λοιπόν να συλλέξουμε τέτοια στοιχεία και όλα τα κράτη-μέλη συλλέγουν τέτοια στοιχεία για τους αλλοδαπούς μαχητές. Αν λοιπόν είναι κάτι σημαντικό για τις μυστικές υπηρεσίες είναι να προστατεύσουν τις πηγές τους γιατί αν υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρα πολύ απλά θα τρομάξουν. Και πάντα μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι χρειάζεται να εξηγήσουμε τα πάντα. Να είμαστε διαφανείς για τα πάντα. Αν πρέπει να σας πούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί το PNR και πώς ε, θα εφαρμοστούν τα κριτήρια στο PNR, ο κόσμος ε, τον οποίο παρακολουθούμε θα αλλάξει τη συμπεριφορά του. Ο επικεφαλής του MI5 για παράδειγμα είπε ότι υπήρξε μία συμπεριφορά από πλευρά του Snowden γιατί πολύ απλά κατάλαβαν πώς παρακολουθούνταν. Αυτό είτε μας αρέσει είτε όχι είναι έτσι για την ιδιωτική σφαίρα. Πέρασα ένα χρόνο για να καταρτήσω το άρθρο 7 και 8 του σχετικού χάρτη, της σχετικής χάρτας. Πρέπει να βρούμε λοιπόν ε, μια ισορροπία Και καλά κάνουμε και φτιάχνουμε ένα στεναρό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων, αλλά είναι υπερβολικά στεναρό, υπερβολικά αποδοτικό και δεν επιτρέψει την ανταλλαγή δεδομένων, δεν θα λειτουργήσει στο νέο πλαίσιο. Άρα θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Εκεί που συμφωνώ είναι ότι υπάρχει έλλειψη οράματος για, την δεύτερη, για τους μηχανισμούς συλλογής και κοινής ε, χορήγηση στοιχείων και δεδομένων. Και στο παρελθόν λοιπόν υπήρχαν τόσο πολλά διαφορετικά συστήματα που αναγκαστικά έπρεπε να υπάρξει μια εναρμόνιση. Υπάρχει μια έλλειψη λοιπόν κοινής, κοινού οράματος, κοινή διαμόρφωσης και αυτό θα αποτελέσει μια πρόκληση για το μέλλον. Το πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε μια καλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων των μηχανισμών αυτών. Τι είδου δεδομένα χρειαζόμαστε. Εγώ Πιστεύω και το επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται να συλλέγουμε στοιχεία και δεδομένα PNR ακόμα και αν ε, στις επιθέσεις ε, στο Παρίσι ο κόσμος πήρε το αυτοκίνητο, οι τρομοκράτες. Ε, μα δεν είναι αυτό επιχείρημα, τι δηλαδή μόνο αυτό το τελευταίο παίρνουμε υπόψη. Τώρα, για να απαντήσω στις άλλες ερωτήσεις. Στην παρούσα κατάσταση το θέμα δεν τίθεται γιατί ε, μας υποχρεώνουν οι υπάρχουσες συνθήκες. Οι συνθήκες όμως λένε κάτι στο άρθρο 4 ότι η εθνική ασφάλεια είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Στο άρθρο 73 όμως λέει ότι τίποτα δεν εμποδίζει τις χώρες μέλη να ενδυναμώσουν την τη συνεργασία μεταξύ των ε, υπηρεσιών πληροφοριών. Και αυτό ακριβώς ζητήθηκε από τις ίδιες ε, τις υπηρεσίες, το CTG, το GATT, να ενδυναμωθεί αυτή η συνεργασία. Αυτό είναι κάτι που γίνεται και αυτό είναι το μήνυμα που εγώ στέλνω. Είναι σημαντικό εκτός του θεσμικού πλαισίου της Ένωσης να διαρθρωθεί πολύ περισσότερο η ε, συνεργασία τους σε επίπεδο πληροφορικών συστημάτων, μονίμων δομών κτλ. Δηλαδή πέρασαν από τη, βιομηχανική συνεργασία από την βιοτεχνική εκτός των θεσμικών πλαισίων της, ε, των συνθηκών. Το θέμα είναι να βρούμε ένα καλό σημείο διασύνδεσης με τις όλες δομές ε, της ε, συνθήκης. Κατά την άποψή μου η Europol θα παίξει καθοριστικό ρόλο, αλλά νομίζω ότι λανθασμένα είναι, θεωρείται μια αστυνομική πλατφόρμα. Για μένα είναι μια πλατφόρμα διασύνδεσης. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να τη βλέπουμε. Θα πρέπει να είναι ένας χώρος ανάλυσης και επεξεργασίας των πληροφοριών. Και για τους ξένους μαχητές βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει μία και μοναδική πλατφόρμα ε, η οποία θα συνεργάζεται και με τα άλλα συστήματα. Τώρα, το δεύτερο ε, ερώτημα. Το θέμα και πάλι αφορά την Europol. Είναι ανώφελο, κατά περίσταση, να απευθυνόμαστε στο ACS. Το τρίτο σημείο. Σύμφωνο ότι πράγματι ε, το συμπλήρωμα του PNR είναι υποχρεωτική χρήση του SIS. Ο κύριος Λόπες αναφέρθηκε στο θέμα του blame gain, της επίρρηψης ευθυνών. Δεν ακούσαμε τις επικρίσεις της Επιτροπής λίπες στο Συμβούλιο. Ενδεχομένως θα μπορούσατε να ενημερωθείτε ότι ήμουν ο πρώτος που αναγνώρισε ότι υπάρχει ανάγκη άμεσης εφαρμογή των όσων αποφασίστηκαν προηγουμένω. και οι Υπουργοί αναγνώρισαν ότι τα είχαν ξαναδεί αυτά τα συμπεράσματα το Φεβρουάριο και ενδεχομένω και πριν το Φεβρουάριο. Πιστεύω λοιπόν ότι συλλογικά υπάρχει αναγνώριση ότι όταν κάτι αναγνωρίζεται στι Βρυξέλλες μετά θα πρέπει να εφαρμόζεται στι χώρε μέλη. Και η Προεδρία και εγώ ο ίδιος θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε αυτή τη δύσκολη συζήτηση την ε, Παρασκευή. Μερικές φορές θα πρέπει να φέρουμε αντιμέτωπους ε, τους υπουργού ε, με δυσάρεστες αλήθειες. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμβεί αυτό, αλλά δεν έχω δει να γίνεται κάποια κριτική από πλευρά της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Είναι αλήθεια ότι για να το πούμε με τον πιο απλό τρόπο, υπήρχε μια βραδίτη, υπήρχε μια βραδίτητα. Δεν θέλω να επιμείνω, αλλά αν δεν έχουμε ένα νέο PNR θα έχουμε εθνικά PNR. Ε, οι χώρες πιστεύουν ότι είναι χρήσιμο. Και νομίζω ότι θα είναι λιγότερο προστατευτικό, λιγότερο ευρωπαϊκό, λιγότερο αποτελεσματικό. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να ξεκινήσουν αυτέ οι διαπραγματεύσει, οι οποίε με βρίσκουν απολύτω σύμφωνο. Τώρα, το ερώτημα. Ε, σχετικά με τη θέση μου, ναι, βεβαίω. Το καταλαβαίνω. Περίεργη λειτουργία, εξ ονόματος ποιου μιλάω. Η θέση μου δημιουργήθηκε από τους επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων και εγώ προσπαθώ να τα φέρω όλα αυτά εις πέρας με τον καλύτερο τρόπο. Μιλάμε για κάτι ιδιαίτερα πολύπλοκο, ένα πολύπλοκο παιχνίδι με πολλούς παίκτες. Προσπαθώ να έχω μια επικοδομητική συμπεριφορά Ενδεχομένω οι διαθέσιμοι πόροι θα μπορούσαν να επεκταθούν. Το θέμα όμω δεν είναι αυτό. Το θέμα μου είναι να συνεργαστώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναπτύξω τι καλύτερε δυνατέ σχέσει για να μπορέσω να κινητοποιήσω του υπάρχοντε πόρου και να εγκαθιδρύσω μια σχέση εμπιστοσύνη έτσι ώστε να μπορώ να ενημερώνομαι για τι ανάγκε του και να τι θέτω σε ένα νέο πλαίσιο. Σε ό,τι φορά το Κοινοβούλιο πάντοτε σα ενημερώνω Ε, προσπαθώ να το κάνω το συντομότερο δυνατόν, προσπαθώ να είμαι έντιμο στις αξιολογήσεις μου. Τώρα, συμφωνώ με αυτό που είπε ο Ραούλ, μιλάμε για ένα καινούριο τομέα για όλους μας. Αναφερόμουν τους Γάλλους γιατί οι Γάλλοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Πριν από τρία-τέσσερα χρόνια η γαλλική κυβέρνηση δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για αυτό το θέμα. Αφορούσε περισσότερο τους Βρετανούς. Οι Βρετανοί έκαναν λάθη αλλά έκαναν και πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις και αυτό επηρέασε το χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών των Δανών, των Γερμανών για παράδειγμα. Και πιστεύω ότι τώρα υπάρχει ανάληψη υποχρέωση από τις περισσότερες χώρες μέλη για να κάνουν κάτι περισσότερο. Και οι Αμερικανοί, και οι Αμερικανοί πριν από μερικά χρόνια δεν είχαν είδηση για αυτά τα θέματα. Τώρα οργάνωσαν μια παγκόσμια διάσκεψη στη Νέα Υόρκη και αυτό σηματοδότησε μια πρόοδο. Είναι πολύπλοκα τα πράγματα. Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να πω ότι έχω ανάμεικτα συναισθήματα συστήματα σε ό,τι αφορά το ρόλο της ιδεολογίας. Μπορεί κανείς να βάλει δύο-τρεις εμπειρογνώμονες να συζητήσουν και ε, δεν θα μπορέσουν να καθορίσουν το πρόβλημα. Ε, τι να πω, έλλειψη στόχου, αποθυμένα για την έλλειψη ενσωμάτωσης, τι θα πω, η ιδεολογία είναι ένας καθοριστικός παράγοντας, αλλά σε τελευταία ανάλυση αυτή είναι μία ε, ε, λύση μαύρο-άσπρο σε ό,τι αφορά τη βίαιη συμπεριφορά. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ είμαι υπέρ της ιδέας του να τα επεξεργαστούμε όλα αυτά. Πολλά ακόμα μπορούμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά το ίντερνετ. Ε, Έχουμε να κάνουμε πολλά με τους ημάμις της Τεχεράνης ε, θα πρέπει να ελέγξουμε τα κέντρα ε. Το θέμα είναι να ζητήσουμε από την Επιτροπή να κάνει περισσότερα, περισσότερα στο θέμα της συνοχής, της καταπολέμησης, της Ισλαμοφομίας, της δημιουργικής σκέψης, της κουλτούρας, της Ισλαμοφοβίας. Υπάρχουν περισσότερα που μπορούμε να κάνουμε στο υπάρχουν πρόβλημα, πρόγραμμα. Ε, κοιτάξτε, το Ευρωπαϊκό Ισλάμ υπάρχουν 20 εκατομμύρια εκατομμύρια μουσουλμάνοι στην Ευρώπη. Ο αριθμός τους θα αυξηθεί. Θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να φτιάξουν μία θρησκεία που να έχει την ίδια βάση με τις άλλες θρησκείες. Ανοιχτή, χαλαρή, συμβατή με τις ευρωπαϊκές αξίες. Και το τίθεται το θέμα της εξωτερικής χρηματοδότησης από μερικέ χώρε μέλη. Αυτή είναι μια δύσκολη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να διεξαχθεί και να διεξαχθεί σύντομα. Υπάρχουν και πολλά άλλα ερωτήματα για την Τουρκία. Για παράδειγμα, ναι, η Τουρκία όλο και περισσότερο ε, έχει εμπλοκή στην καταπολέμηση του ISIS, το είδαμε στην ε, Άγκυρα και αυτά είναι καλά νέα θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Υπάρχουν ε, βεβαίως και πολλά άρα θέματα και πολλές άρες Σε ό,τι αφορά όμως την αντιτροποκρατία νομίζω ότι έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος. Θα πρέπει όμως να αναλάβουμε δέσμευση ε, νομίζω ότι με το να είμαστε απλοί παρατηρητές δεν θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε τα πράγματα. Όσο μεγαλύτερη εμπλοκή έχουμε τόσο περισσότερο θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην εξέλιξη των πραγμάτων και στη βελτίωση της ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα λοιπόν... Ε, ε ξέρω ότι δεν ήταν να απαντήσετε σε όλε τι ερωτήσει, αλλά σα ευχαριστώ που προσπαθήσατε τουλάχιστον να απαντήσετε σε πιο πολλέ εξ αυτών. Όλοι Ολιβιέ, θα αναγκαστώ να σου ζητήσω να είσαι σύντομο, ε, γιατί έχει περάσει πολύ η ώρα. Πέντε λεπτά, μάλιστα, επιγραμματικά. Αρχικά δεν θέλω να πω ότι ε, ζούμε βεβαιασμένα είναι σαφές ότι επιταχύνουμε τις ενέργειές μας μετά τις δημοκρατικές επιθέσεις και όπως ε, ο Φούρναρης πρέπει και εμείς να δουλέψουμε μέσα τη νύχτα για να έχουμε φρέσκο ψωμί το πρωί. Αυτό γίνεται και στην Κομισιόν αυτή τη στιγμή. Όμως υπενθυμίζω ότι εδώ και 10 χρόνια έχουμε ευρωπαϊκή στρατηγική καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, που βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες και συνδέεται και με τη σημερινή συζήτηση, πρόληψη, προστασία, δίωξη και ανταπόκριση εργαζόμαστε κάποιες φορές ε, ατύπως ε, και με τις ε, υπηρεσίες, μυστικές υπηρεσίες των κρατών μελών στο σύνολο αυτών των τεσσάρων πυλώνων. Όσα προτείνουμε και όσα κάνουμε ανταποκρίνονται συγκεκριμένα κριτήρια και ελέγχους. Όλες μας οι προτάσεις ανταποκρίνονται σε αυτό το τετραπλό τεστ της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας, τη ε, τήρηση των θεμελιώδων δικαιωμάτων κτλ. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εξετάζει όλα αυτά. Οι υπηρεσίε τη, η νομική υπηρεσία τη Κομισιόν, που ελέγχει ακριβώς ε, την ορθότητα των πράξεών μα. Για την μη υλοποίηση, πράγματι επιβεβαιώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα που η μεταβατική περίοδος των 5 ετών της Συνθήκης Λισαβόνα έχει περάσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει πλήρω ευθύνε τη ε, ό,τι αφορά τη διαδικασία τη Και κάποιε μάλιστα ετοιμάζονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα αποτελέσει θεματοφύλακα τη συνθήκη ε, στο μέγιστο βαθμό που τη αναλογεί. Να σα δώσω μερικά παραδείγματα μη εφαρμογή τη νομοθεσία. Όταν λέμε μη εφαρμογή, γνωρίζουμε ότι κάτι έχει προταθεί, κάτι έχει αποφασιστεί ή νομικό ή σε πρακτικό πλαίσιο και απλώς δεν εφαρμόζεται. Ο λόγος μπορεί, οι αιτίες μάλλον μπορεί να είναι πολλές. Έλλειψη πολιτικής βούλησης, τεχνικές ασυμβατότητες, έλλειψη πόρων και ο Ζήλ αναφέρθηκε σε ε, παροχημένα πληροφορικά συστήματα στα σύνορα. Πολλές είναι οι αιτίες. Δύο παραδείγματα. Η Europol τώρα προσπαθεί να διασυνδεθεί και με τα 28 κράτη-μέλη ε, για την ανταλλαγή πληροφοριών να πάμε σε επίπεδο εμπιστευτικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια κράτη-μέλη ούτε καν ζήτησαν τη σύνδεση. Αν λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε για ανταλλαγή με πληροφοριών με προστατευμένο τρόπο, πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρξει γραμμή. Είναι δωρεάν. Η Europol θα το κάνει για εσά. Αν δεν το ζητάει κανεί, υπάρχει θέμα. Δεύτερον, το σημείο εστίασης της Europol στους ε, ταξιδιώτες. Περίπου 5.000 ε, αλλοδαποί μαχητές ευρωπαϊκής καταγωγής στη Συρία και στο, και στο Ιράκ. Ε, συνολικά 20.000 από 100 χώρες. Εμείς έχουμε μόνο 1.500 ονόματα είναι πολύ μεγάλο το χάσμα λοιπόν. Και δυστυχώς ορισμένες ε, χώρες έχουν δώσει περισσότερα στοιχεία από ό,τι τα δικά μας τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης και δέσμευσης. Τώρα για την ανταλλαγή πληροφοριών. Έχουν υποθεί πολλά. Ξέρουμε τα όσα αναφέρει η συνθήκη. Είναι κάτι άλλο σημαντικό που ήθελα να θίξω. Πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν σημαντικέ διαφορές μεταξύ μυστικών πληροφοριών, αρχών επιβολής του νόμου, αστυνομία δικαστικών αρχών. Από πλευράς εντολής, ε, τεχνικών έρευνας, συστημάτων εποπτεία και γενικών στόχων. Η συλλογή πληροφοριών ή μυστικών πληροφοριών δεν υπόκειται στους ίδιους κανόνες, αρχές, ε, ε, κανόνες εποπτείας, και παρακολούθησης, όπως είναι οι κλασικές μέθοδοι αρχών επιβολής του νόμου. Αυτό υπάρχει στα κράτη-μέλη. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κενό που προσπαθούσε να συμφιλειώσει και ο Ζιλ παρουσιάζοντας τη Europol ως τον ε, κεντρικό πυρήνα, αν θέλετε. Αυτό είναι ένας τρόπος, αλλά αυτή η διαφοροποίηση υπάρχει παντού και στα κρατημέλη. Υπάρχουν λύσεις, ναι. Υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας, ναι σε συγκεκριμένα ζητήματα. Χωρίς ανταλλαγή επιχειρησιακών δεδομένων, αλλά στο επίπεδό μας, στρατηγικά, ναι. Γι' αυτό και δίνουμε ε, αξιολόγηση κινδύνου στις άλλες γενικές διευθύνσεις. για να προσδιορίσουμε τον κίνδυνο σε ένα συγκεκριμένο τομέα, σε συγκεκριμένο μότο operandi. Και μετά ο καθένας ε, παίρνει τις αποφάσεις του. Ο Ζιλ ανέφερε τις εργασίες μας ό,τι αφορά την ε, πολιτική αεροπορία και την προστασία σε αυτό το επίπεδο. Πράγματι λοιπόν ε, υπάρχει δυνατότητα πρακτικής συνεργασίας, όμως είναι μια αργή διαδικασία οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και αυτό κάνουμε ενώ περιμένουμε τις αποφάσεις σε ψηλότερο επίπεδο για τις πρόδρομες ε, ύλες, το CBRN και τα σχέδια δράσης για τις εκρηκτικές ύλες. Πράγματι, το 2008 είχαμε ένα σχέδιο δράσης για το CBRN. Είχαμε και το 2009 σχέδιο δράσης για τις εκρηκτικές ύλες. Όλες οι δράσεις, σχεδόν όλες οι δράσεις, έχουν υλοποιηθεί. Εγώ αναφέρθηκα συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις πρόδρομες ύλες και ουσίες. Ήταν και στο πρόγραμμα της Κομισιόν 2016. Στα μέσα της χρονιάς θα επανέλθουμε μια αναθεωρημένη στρατηγική για τα CBRN. Χθε ήμουν στο Μπορσέτ, το κτίριο κοντά εδώ, και προείδρευσα μια συνάντηση σε πραγματικά ειδικών σε ζητήματα ε, ε βομβών, σε ό,τι αφορά τις ε, dirty bombs όπως αποκαλούνται, συγκεκριμένες πρακτικές εντοπίσαμε, θα υποβάλουμε εκθέσεις για να δούμε πού μπορεί να σημειωθεί η πρόοδος, πού υπάρχουν κενά και το καθεξής. Για το ζήτημα των ανθρωπιστικών επιστημών, συμφωνώ απολύτως μαζί σα ότι για να δημιουργήσουμε ένα εναλλακτικό αφήγημα ε, και να δώσουμε αντίστοιχη φωνή και σε άλλες ε, απόψεις, πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τα υποφόσκοντα φαινόμενα, γιατί αν, αν δεν εντοπίσουμε τις αιτίε, δεν θα εντοπίσουμε και τη λύση. Γι' αυτό το φόρουμ IT και το δίκτυο RAN είναι τόσο σημαντικό. Εδώ πέρα και το κέντρο αριστείας θα πρέπει να περάσει από ανάλυση Συγκεκριμένε αναλύσει λοιπόν, εξέταση βέλτιση πρακτικών με σημεία επαφή και το καθεξή. Θέλουμε να δούμε τι γίνεται στη Δανία, τι γίνεται στη Βαρκελόνη. Να μπορεί κάποιο ε, να τηλεφωνήσει, ε, σε εκείνο, να πάρει τηλέφωνο και το μέλο και να δει. Και μετά πρέπει να περάσουμε στη δράση. Αυτό έκαναν. Και τώρα κινούνται με τη στήριξή μα και παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτική ε, και προ κράτη-μέλη και τρίτες χώρε. δεν ξέρω, είπατε για τον Ιανουάριο. Εγώ νομίζω ότι τα τελευταία κονδύλια του ΡΑΝ τα ταπανίσαμε τον περασμένο Σεπτέμβρη. Το τελευταίο εργαστήριο έγινε ακριβώ ε, για τα πληροφορικά συστήματα. Εν τω μεταξύ, ακολουθήσαμε την ε, διαδικασία διαλογή ε, για το κέντρο αριστεία ΡΑΝ, αλλά ο προηγούμενο συμβασιούχο δούλεψε μέχρι και το Σεπτέμβρη αν έρθετε σε επαφή μαζί τους θα σας δείξουν τους συμμετέχοντες, τα πρακτικά, τους στόχους και το καθεξής. Και τα τελευταία δύο, εν συντομία, για το ξέπλυμα χρήματος, τι λείπει στην τέταρτη οδηγία. Η οδηγία αυτή βασίζεται σε μια νομική βάση της εσωτερικής αγοράς. Το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος ποινικοποιείται εν μέρη, αλλά μη συστηματικά, σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη. Θεωρούμε χρήσιμο, αλλά αυτό το εξετάζουμε, δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει, συμπληρωματικά, όχι υποκαθιστώντας ε, άλλα στοιχεία, να έχουμε μία ε, οδηγία υπό το 83.1 μόνηση των υφιστάμενων συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κάποια παραθυράκια ε, σε ό,τι αφορά την, ε, το ξέπλυμα χρήματο εξαμελίας, για παράδειγμα. Εδώ υπάρχει κάποια προστιθέμενη αξία. Και στο τελευταίο, να καθησυχάσουμε και του Σουηδούς κυνηγού. Ήθελα απλώ να πω ότι τα πυροβόλα όπλα, εγώ το αντίθετο έλεγα βασικά, δεν ξέρω αν δεν ήμουν σαφή. το πρόβλημά μα είναι η μεγάλη μαύρη αγορά, είτε το παροπλισμένων πυροβόλων όπλων ή η μαύρη αγορά των στρατιωτικών ε, όπλων από είτε καινούριων είτε μεταχειρισμένων από ε, γειτονικέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Όμω θέλουμε να δράσουμε και αναλογικά. Θα δείτε λοιπόν στην οδηγία έχουμε ξεχωριστέ κατηγορίε πυροβόλων όπλων. Κάποια απαγορεύονται εντελώ, κάποια επιτρέπονται ε, υπό την προπόθεση ύπαρξη άδεια, το οποίο ισχύει για του κυνηγού για άλλα χρειάζεται μόνο μία δήλωση και τα, κάποια άλλα θα, ε, θα επιτρέπεται πλήρωση η πώλησή τους. Υπάρχει βεβαίως ε, το πνεύμα της ελεύθερης ε, διακίνησης εμπορευμάτων. Από εκεί ξεκινήσαμε, αλλά τώρα θέλουμε να το περιορίσουμε κάπως, να έχουμε στο νου μας και την ασφάλεια. Αλλά βεβαίως δεν υπάρχει κίνδυνος για τους Σουηδούς κυνηγούς. Απλώ θα υπάρχει ένα εύρωστο στο σύστημα, είτε εκ των προτέρων αδειοδότηση, είτε καταχώρησής του. Ευχαριστούμε πολύ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που απαντήσατε τι ερωτήσει των ε, μελών τη Επιτροπή. Συνάδελφοι, ήταν πάρα πολύ μακριά η συζήτηση και πολύ γεμάτη. Έχουμε ξεπεράσει το όριο που προβλεπόταν και αυτό γι' αυτό εγώ επέτρεψα στους ε, βουλευτέ να μιλήσουν παραπάνω, αλλά Θεωρώ ότι τα θέματα αυτά που βρίσκονται στη φάση τρομερούς διαλόγου είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ελπίζω να το εκτιμούν αυτό οι ομιλητέ. Νομίζω ότι συμπεριληφθήκε η συζήτηση για πολλά βασικά θέματα, ε, θέματα εφαρμογή και υλοποίηση που μα απασχολούν. Άρα θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ μεστή αυτή η συζήτηση και πραγματικά συμμετείχαν σχεδόν όλοι τα μέλη τη Επιτροπή σα. ευχαριστώ πάρα πολύ και του τρει για τον χρόνο που μας αφιερώσατε σήμερα το πρωί. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, σημερινή συζήτηση και ζητώ συγγνώμη στους προσκεκλημένους για τα επόμενα θέματα που περίμεναν. Σας παρακαλώ να φύγετε, αν χρειαστεί να φύγετε, ήσυχα από την αίθουσα. Um, Συνάδελφοι, προσκεκλημένοι μας. Έρχονται στα μπροστινά έδρανα να σας παρουσιάσω ε, την εκθεσία αυτή και το συγγνώμη για όλους τους συναδέλφους, σε όλους τους συναδέλφους που περίμεναν γιατί ξεπεράσαμε το χρονικό όριο. Στο 22, συμφωνία μεταξύ, για τη συνεργασία μεταξύ Γεωργίας και Ουκρανία, το 23 μεταξύ Eurojust και Μαυροβουνίου. Τα ζητήματα λοιπόν αυτά, τα θέματα αυτά θα συζητηθούν από κοινού και καλωσορίζω τον κύριο, την κυρία Μισελ Κόνιγκς, η οποία είναι η πρόεδρος της Eurojust, ε, καταφτάνει, θα μας παρουσιάσει τις δράσεις που έχουν ληφθεί από το σώμα της Eurojust μετά από εξωτερική ανάλυση που έγινε για τη δραστηριότητα της Eurojust και γενικά ε, την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Eurojust. Επίσης, ε, ενδεχομένως να πάρει το λόγο και να πει δύο λόγια για τις δύο συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Eurojust και Ουκρανίας και Μαυροβουνίου. Αντίστοιχα, τις οποίες, ε, για τις οποίες γνωματοδοτεί η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Και στο δεύτερο τμήμα θα πάρουν το λόγο οι δύο αντίστοιχοι εισηγητές για την παρουσίαση του σχεδίου έκταση από την κυρία Κάφμαν. Ζητώ συγγνώμη και στου δύο εισηγητέ για την καθυστέρηση. Και μετά η κυρία Γκρίσπεκ θα πάρει το λόγο, η οποία είναι και η εισηγήτρια για την συνεργασία μεταξύ γύρω Τζάστ και Μαυροβουνίου. Και μετά θα πάρουν το λόγο τα μέλη της Επιτροπής. Ζητώ λοιπόν και πάλι συγγνώμη από όλους τους συναδέλφους που χρειάστηκε να περιμένουν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την κυρία Κόνιγκς. Αν θα μπορούσατε να συμπτύξετε κάπως την παρουσίασή σα για να κερδίσουμε λίγο από το χαμένο χρόνο. Και για τους συζητητές οι οποίοι ενδεχομένω να χρειαστεί να φύγουν λίγο νωρίτερα. Και λυπάμαι που σα πιέζω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μέλη, συγητές της Επιτροπής Λίπεντου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι τιμή και χαρά για μένα να σας μιλήσω για τις δραστηριότητες της Eurojust. Θα ήθελα να δω στην έκθεση Young για την εξωτερική αξιολόγηση της Eurojust. Αυτή είναι μία ανεξάρτητη αξιολόγηση. Διαφάνεις παρακαλώ. Αυτή η αξιολόγηση γίνεται κάθε πέντε χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη τέτοια άσκηση που είχαμε. Το πρόγραμμα δράσης το μεταξύ συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο. Μετά είχαμε την έκθεση της Ernst Young που είναι μια ανεξάρτητη έκθεση που επικεντρώθηκε σε τρία σημεία την εφαρμογή των, αποφασιών της Eurojust, τον τρόπο με τον οποίο η Eurojust με βάση αυτή την κοινή απόφαση ε, ε, βέτυχε τους στόχους της και την αποτελεσματικότητα της Eurojust. Στην έκθεση Ernst Young έγινε μία αναφορά σε όσα πήγαν καλά και βεβαίως υπεγράμμισαν και ορισμένους τομείς αφήνοντας κάποιο περιθώριο για βελτιώσεις. Θα πρέπει να πούμε ότι μερικές από τις συστάσεις αναφέρονται σε μέτρα που δεν θα πρέπει να ληφθούν από την ίδια τη Eurojust. Εμείς θα επικεντρωθούμε κυρίως στη Eurojust και μετά στους άλλους σημαντικούς παίκτες. Σε ό,τι αφορά θέματα λειτουργικά, έγινε μια αξιολόγηση από μέρους των κρατών μελών. Αυτό είναι κάτι κεκτημένο, κάτι που καταφέραμε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι μας είναι περιορισμένοι και η δουλειά που έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ. οι συστάσεις. Οι συστάσεις διατυπώνονται σε οκτώ τομείς. Ο πρώτος τομέας αφορά την ανάγκη του να συνεχίζουμε να διαδιαβατρίζουμε ενεργό ρόλο για να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του 2008 του Συμβουλίου. Υπάρχει μια σημαντική σχέση με την ομάδα εργασία Ζαμπέλ, οι οποίες περάτωσαν, ε, έκαναν την τελική διαμόρφωση της έκθεσης και υιοθετήθηκε ένα πρόγραμμα εργασίας από την Eurojust το 2008. Αυτό ακριβώς κάνουν οι χώρες μέλη σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Να υπάρχει δηλαδή μια σχέση μεταξύ των δύο εκθέσεων. Νομίζω ότι οι εκθέσεις αυτές ήταν την κατάλληλη στιγμή, γιατί και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναπτύξουν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για την περαιτέρω ανάπτυξη της Eurojust και του κανονισμού για την Eurojust. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να δούμε τι λένε οι εξωτερικοί ε, εκτιμητές, τι είπαν οι πελάτες ας πούμε σχετικά με την απόφαση αυτή και γενικά πώς αναπτύσσει τη δράση της η Eurojust. Το Πρώτο σημείο, η πρώτη σειρά από συστάσεις έχουν σχέση με το άρθρο 12 της απόφασης του Συμβουλίου και τα συστήματα εθνικού συντονισμού της Eurojust. Από αυτή την άποψη λάβαμε ορισμένα μέτρα και 2008 Προτίσαμε το ΦΙΣ Σουεντουάζ αυτά. Μπορείτε να βρείτε τα βρείτε των εθνικών αντιπροσώπων στο extranet της Eurojust. Όλα αυτά τα επικαιροποιούμε μία φορά το χρόνο και έτσι γνωρίζουμε σε τι σημείο ε, βρίσκεται η εφαρμογή του ENCS. Οργανώνουμε και τακτικές συναντήσεις, έγινε μια συνάντηση το 12, το 14 και θα γίνει και μια άλλη το Φεβρουάριο του 16 σε μια προσπάθεια να συναντηθούν όλοι αυτοί οι εμπειρογνώμονες για να δουν πώς μπορούν να συνεργαστούν στα πλαίσια του ENCS. Επίσης, οργανώνονται συναντήσεις μεταξύ της Eurodust και του EGN μεταξύ των τεστ τη ε, ε, Eurojust και των σημείων, εθνικών σημείων επαφή έτσι ώστε η Eurojust να λάβει καλύτερη γνώση των πραγμάτων και να υπάρχει και μία αλληλεπίδραση. Η Eurojust από την άλλη προωθεί την εμπλοκή των μελών του ENCS σε διάφορα σεμινάρια ε, marketing Πηγαίνουμε στις χώρες μέλη για να ενημερώσουμε τους πελάτες πώς θα μπορούσαν να κάνουν μια καλύτερη χρήση των υπηρεσιών και προγραμματίζουμε να, το, να οργανώνουμε τακτικές ε, τέτοιες συνεδριάσεις για να μπορούμε να εστιάζουμε συγκεκριμένα θέματα. Αυτό αποκοινούμε τα μέλη του ENCS για να μπορούμε να διοχετεύουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες. Μετά ένα τεχνικό θέμα. Λαμβάνουμε υπόψη μας το πώς τα μέλη θα μπορούσαν να έχουν σχέση στο σύστημα διαχείρισης της Eurojust. Yeah, I want to continue. How many, how many seconds do I have? Maybe another, how long were you thinking? Another five minutes? Uh, five, five minutes? We'll, we'll do. Good. Άλλα πέντε λεπτά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και αυτό λοιπόν έχει να κάνει και με τις ασφαλείς συνδέσεις. Έχουμε 14 ασφαλείς συνδέσεις στην παρούσα φάση, έχουμε 28 κράτη-μέλη και αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνουμε πιο πολλές προσπάθειες στα κράτη-μέλη για να δούμε σε τι βαθμό μπορούν να συνδεθούν μαζί μας. Με τη γραμμή λοιπόν αυτή, στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε ότι υπάρχει το άρθρο 13 για τις πληροφορίες που θα πρέπει να χορηγούνται στην Eurojust Επίσης και εδώ συνεργαζόμαστε για να υπάρχει ένας εύκολος τρόπος ενημέρωσης της Eurojust για το τι είδους διασυνοριακές έρευνες θα πρέπει να γνωρίζει για ποιε τέτοιε έρευνε θα πρέπει να είναι ενήμερη η Eurojust υπό το άρθρο 30ε, το οποίο λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να δίνουμε και feedback στα κράτη-μέλη, παρά το γεγονός ότι έχουμε λάβει κάποια βήματα για να υπάρχει ενημέρωση των εθνικών αρχών και για να υπάρχει και μια εναρμονισμένη ε, προσέγγιση στην διαχείριση δεδομένων της Eurojust. Το 2014 έχουμε εγκρίνει μια γενική πολιτική η οποία έχει και μπει στο γενικότερο σύστημα. Και τέλος προγραμματίζουμε ένα ετήσιο μηχανισμό feedback για τα κράτη-μέλη για τις εκθέσεις αναχώρας. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Είναι μια ετήσια έκθεση, αναεθνική ανα υπηρεσία για τις λειτουργικές ε, επιχειρήσεις. Συστάση υπαριθμό 1. Σύσταση υπαριθμό 1. Μετά την εφαρμογή του, της απόφασης του Συμβουλίου. Κοιτάξτε, έχει εφαρμοστεί, αλλά όχι με ενθουσιασμό χρησιμοποιείται για να έρχονται σε επαφή μαζί μας νύχτα και μέρα μέσω κινητών τηλεφώνων. Αλλά αυτό το σύστημα έχει χρησιμοποιηθεί μόνο περιστασιακά, με επιτυχία βέβαια. Εφαρμογή με σε πραγματικό χρόνο και το καθεξής. Έχει χρησιμοποιηθεί λοιπόν με επιτυχία, αλλά όχι συστηματικά, όχι ενθουσιοδός. Δεύτερη σύσταση. Σε σχέση με την εφαρμογή της στρατηγικού σχεδιασμού, θέτοντας ε, κάποιες προτεραιότητες να κινητοποιηθούν οι σχετικές ε, τα σχετικά μέσα για να υπάρχουν λοιπόν αυτές οι προτεραιότητες να μπορούν να υλοποιηθούν. Λαμβάνουμε λοιπόν διαφόρων ειδών ετήματα αλλά έχουμε και την ατζέντα ιστορικής ασφάλειας, έχουμε και την μεταναστευτική ατζέντα από την αρχή του έτους και για τα επόμενα πέντε χρόνια θα αποτελέσουν τις πλέον ε, κορυφαίες προτεραιότητες όπως είναι και η τρομοκρατία, το κυβερνοέγκλημα. Εστιαζόμαστε λοιπόν σε στρατηγικούς τομείς για να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους και να δούμε μετά την αποδοχή των προτεραιοτήτων, πώς μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε. Η τρίτη σύσταση τώρα. Πιστεύουμε ότι ο νομοθέτης θα πρέπει να ορίζει καλύτερα τους ρόλους που διαδραματίζουν οι διάφοροι φορείς και αυτό αποτελεί μία ερμηνεία του Συμβουλίου. Ποιος είναι ο, ο ρόλος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του καθεξής και του Σώματος. Φυσικά δεν μπορούν να αλλάζουν συνέχεια οι μέθοδοι εργασία, αλλά θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικές. Να υπάρχει μια εκτελεστική επιτροπή, για παράδειγμα, η οποία θα έχει πιο πολλέ τέτοιε και θα τι εκχωρεί αναλόγω. Αυτό είναι μια δικασία υπό εξέλιξη, αλλά θα ε, περιληφθεί και στον κανονισμό. Άρα αυτό θα αποτελέσει έργο του νομοθέτη. Σύσταση υπαριθμών 4. Εναρμόνιση των εσωτερικών δομών. Έχουμε ομάδες, ομάδες εργασίας, ε, task forces. Ε. Θα θέλαμε λοιπόν να επικεντρωνόμαστε πιο πολύ σε συγκεκριμένα έργα, με ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, με σαφή λογοδοσία και αποτελέσματα τα οποία παρακολουθούνται. Ουσιαστικά αυτό συνδέεται με την σύσταση παριθμών 2 για τις στρατηγικές προτεραιότητες, η πέμπτη σύσταση. Πιστεύουμε ότι η κανόνες θα πρέπει να εναρμονίζονται και να είναι πιο συνεπείς, ε, γιατί αυτό επηρεάζει και την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. 28 είναι τα κράτη-μέλη, 28 είναι και οι εθνικές υπηρεσίες, 30 διαφορετικές λοιπόν ε, νοοτροπίες και το θέμα λοιπόν είναι να υπάρξει εναρμόνιση όλων των τρόπων εργασία, των δεσμευτικών και μη δεσμευτικών κανόνων. Αυτό είναι υπό εξέλιξη, πολλά έχουμε κάνει προς την κατεύθυνση αυτή, θα αποφασίσουμε από αυτών των θεμάτων. Το πρώτο τρίμηνο το 2016 για τις ε, προηγούμενες συστάσεις, θα ήθελα να πω το εξής. Προβλέπονται συναντήσεις για να ληφθούν αποφάσεις για όλα τα θέματα αυτά, τα οποία παρακολουθούνται ως τώρα. Είστε σας είπα μόνο έξι. Επόμενη διαφάνεια πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, μια εναρμονισμένη διαδικασία και στις εθνικές υπηρεσίες, προκειμένου να είναι η πραγματική η αρρωγή από πλευρά ε, των αρχών. Έχουμε καταρτήσει ένα εγχειρίδιο για τις ε, δράσεις αυτές, το οποίο και θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλη του χρόνου για διάφορους όρους και τρόπους εργασίας, ε, και μιλάμε για την Ευρώπη που είναι κάτι παραπάνω από το άτρισμα των 28 διαφορετικών διαδικασιών. Έβδομη σύσταση και τελευταία. Οι αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες προκειμένου να έχουν καλύτερη αποδοτικότητα μέσω πιο εναρμονισμένων και εφαρμοσμένων τρόπων εργασίας. Η Eurojust λοιπόν εργάζεται εδώ πέρα για την κατάρτιση δικτών για να προσμετρούνται τα αποτελέσματα των στόχων και να υπάρχει και ένα πιο συνεπές και συνεκτικό σύστημα παρακολούθησης το 2016. Ξέρουμε λοιπόν που είναι η στρατηγική τομή και θα πρέπει να κάνουμε την ίδια άσκηση και για τις εκτελεστικές πτυχές στοιχείο υπαριθμών 8. Σύσταση υπαριθμών 8. Να συνεχίσουμε να παίζουμε ενεργό ρόλο για την ε, εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και να συνεχίσουν ε, να υποστηρίζονται οι σχετικέ δραστηριότητε των οργανώσεων. Και αυτά λοιπόν συνδέονται με τις υπόλοιπε δραστηριότητε. Ευχαριστούμε πολύ, Μισελ. Να δώσουμε τώρα το λόγο ε, στους ε, εισηγητές. Σιλβιά. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, σας ευχαριστώ κυρία Κόνη. Εκτενέστατη η παρουσίασή σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν τη σημερινή συνεδρίαση, κοίταξα την, την ε, των Ernst Young με μεγάλο ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο για την υπερτερά εξέλιξη της Eurojust, όπως είπατε και εσείς. Πρωτού που για τη συμφωνία με την Ουκρανία, θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση. Αυτό παίζει και στην αξιολόγηση του Ernest Young ρόλο, αλλά και στη δική σας παρουσίαση. Εξακολουθούν να υπήρξαν προβλήματα, από ό,τι φαίνεται, στην ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη-μέλη. Ίσως θα μπορούσατε να μας περιγράψετε ποια είναι τα βασικά προβλήματα. Γιατί αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών εξακολουθεί να είναι ελλειπής, να μην είναι όπως θα θέλαμε. Για τη συμφωνία με την Ουκρανία, κύριε Πρόεδρε, δεδομένης και της χρονικής πίεσης, θα κάνουμε μερικές περιορισμένες παρατηρήσεις. Πρόκειται για μια συμφωνία σύνδεσης μεταξύ Eurojust και Ουκρανίας, σε συνεργασία και σε σύνδεση για την καταπολέμηση σοβαρών εγκληματικών πράξεων, του οργανωμένου ε, εγκλήματο και τη τρομοκρατία συγκεκριμένα. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει διατάξει για την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ Eurojust και Ουκρανία. Για παράδειγμα, ε, η απόσπαση συνδέσμων, ανταλλαγή πληροφοριών και το καθεξής. Και αυτό που μας φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό είναι η κοινή η υπηρεσία ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 26 της απόφασης ε, της Eurojust. Συμφώνησε η Eurojust λοιπόν προς ε, την κατευθυνσία αυτή και ότι αυτή η υπηρεσία διαπίστωσε ότι όλες οι προτάσεις που υπέβαλε η Eurojust για τη συμφωνία αυτή έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία και το θέμα της προστασίας των δεδομένων ρυθμίζεται με σαφήνεια. Η Ουκρανία είναι από το 81 μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει εξασφαλίσει ότι υπάρχει ανεξαρτησία για την προστασία των δεδομένων. Αυτό κατοχυρώνεται και από το Σύνταγμα της Ουκρανίας. Συνολικά λοιπόν πιστεύω ότι έχουμε πλέον μια καλή συμφωνία μπροστά μας και ότι το, Συμβου... το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να εγκρίνει τη συμφωνία αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η Νάταλη τώρα είναι η συγγήτρια για τη συνεργασία μεταξύ Eurojust και Μαυροβουνίου. Ευχαριστώ, Κλοντ. Ευχαριστώ και την κυρία Πρόεδρο για τι εξηγήσει τη ε, και τι παρατηρήσει τη Eurojust για το επόμενο διάστημα. Θα είμαι σύντομη, παρότι έχουμε και λίγο χρόνο στη θέση Μα χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να εξετάσουμε και αυτό το φάκελο. Θα ήθελα να επενθυμίσω μόνο στου αδέλφου ότι Βάσει της συνθήκης ε, ε, υπάρχει μόνο διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, δεν υπάρχει συναπόφαση δηλαδή. Επομένω, ε, δεν υπάρχει πραγματική δυνατότητα τροποποίηση των συμφωνιών. Μπορούμε απλώ να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μα ή να την αρνηθούμε. Ταυτόχρονα πρέπει να υπενθυμίσουμε κυρία Πρόεδρε ότι τα τελευταία χρόνια Eurojust ε, συνεχώς αναπτύσσεται και πλέον ε, αποτελεί ένα από τους κεντρικούς ε, φορείς δικαστικής συνεργασίας σε ποινικά ζητήματα. Ταυτόχρονα έχουμε και την και νέα δυνατότητα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο, εξάρθρωση ε, κυκλωμάτων οργανωμένου εγκλήματο και αυτό μα βοήθησε να κατανοήσουμε ότι μία αποτελεσματική συνεργασία και μία κοινή συντονισμένη απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ένα απαραίτητο στοιχείο. Από αυτή την άποψη λοιπόν ο ρόλος ε, του οργανισμού για την βελτίωση της συνεργασίας είναι και σημασία στοιχεία, όπως και εσείς υπενθυμίσατε. Και υπό το φως ε, των ε, τρομοκρατικών επιθέσεων πριν από μερικές μέρες στη χώρα μου. Τελικά, συνάδελφοι, νομίζω ότι οι άνθρωποι που επλήγησαν από αυτές τις ε, τρομοκρατικές επιθέσεις ε, στο Παρίσι δεν περίμεναν αυτή τη δημόσια συζήτηση. Νομίζω ότι έτσι συμβάλλουμε ε, περισσότερο στην απώλεια αυτής της λίγης αξιοπιστίας που έχει απομείνει στην Ευρώπη. Το μέλλον είναι το παρόν. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει ε, η Ευρώπη για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα αυτών των ανθρώπων. Γιατί αν δούμε ότι το υφιστάμενο πλαίσιο δεν επιτρέπει να υλοποιηθούν κάποια απαραίτητα στοιχεία, τότε θα πρέπει να το τροποποιήσουμε και να έχουμε αποτελέσματα σε μικρό χρονικό διάστημα. Το οργανωμένο έγκλημα Κάθε μέρα βλέπουμε ότι και η τρομοκρατία, η απάτη, η διαφορά δεν έχουν σύνορα. Κάθε μέρα όχι μόνο βλέπουμε, αλλά εφιστάμεθα για τις συνέπειες ε, αυτής ε, της εγκληματικής ενέργειας, εγκληματικής, τρομοκρατικής ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει σύνορα αυτή η δραστηριότητα και έτσι ούτε η δική μας ανταπόκριση πρέπει να έχει σύνορα. Και αν θέλουμε μια διακυβερνητική συνεργασία θα πρέπει να είναι και δυναμική και αποτελεσματική. Και γι' αυτό θα πρέπει να διευκολύνουμε τις ε, διαδικασίες ε, έρευνας και αυτό θα πρέπει να ιεραρχηθεί ως προτεραιότητα. Αυτές οι συμφωνίες είναι κλασικές, ε, σχεδόν ταυτόσιμες ό,τι αφορά το περιεχόμενό τους και αντίστοιχες και με συμφωνίες που έχουν συναυθεί ε, με τους στόχους ενίσχυσης της συνεργασίας, ε, διορισμού ε, δικαστικού συνδέσμου, σημείων επαφής και το καθεξής. Και όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, δεν νομίζω ότι δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα. Και γι' αυτό σας καλώ συνάδελφοι να εγκρίνετε αυτή τη συμφωνία. Μερικά όμω σύντομα σχόλια. Πρώτον, ερωτήσεις μάλλον. Θα μπορούσατε κυρία Πρόεδρε να μας ε, αναφέρετε για ποιους λόγους ιεραρχήσατε αυτές τις δύο χώρες ως προτεραιότητες. Είναι οι πάλι κατά του οργανωμένου εγκλήματος στα Βαλκάνια που ξεφεύγει από κάθε όριο. Και γιατί επιλέξατε αυτές τις χώρες και όχι το Κοσμοπέδιο για παράδειγμα ή κάποιο άλλο. Δεύτερον, ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχετε θέσει στο προσκήνιο και ποιες είναι οι χώρες που θεωρούνται χώρες προτεραιότητας για τη Eurojust. Τρίτον, σε σχέση με την έκθεση δραστηριοτήτων ε, του 2013, αναφερθήκατε στην προτεραιότητα που είχε δοθεί στη σύναψη συμφωνίας ε, με τη Ρωσία τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση, υπάρχει πρόοδος, συνεχίζεται, έχει διακοπή, τι συμβαίνει. Πρώτο τελευταίο ερώτημα. Θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενημερώνεται πιο συστηματικά σε σχέση με τις προτεραιότητες σε αυτό το πολύ σημαντικό κλάδο της δικαστικής αστυνομικής μάλλον συνεργασίας με άλλα κάτι μέλη. Και τελευταίο ερώτημα, το οποίο είναι τακτικά αναφέρεται. Ήδη υπάρχει τέτοια, τέτοιες συμφωνίες που δεν έχουν ακόμα τεθεί ε, σε ισχύ. Ποια είναι η αποτελεσματικότητά τους, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για την ωφελημότητά τους ε, και αυτός ο εισαγγελέας σύνδεσμος ε, επίσης είναι χρήσιμος θεσμός. Είναι κάτι το οποίο έχει απτά αποτελέσματα. Θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες γιατί καλό θα ήταν να λάβουμε περισσότερα στοιχεία και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δύο μέλη ζήτησαν το λόγο. Κύριε Στατίνα, κύριε Γκόμες, παρακαλώ. Είναι μεγάλη η τιμή για μένα το ότι έλαβα αυτή την έκθεση. Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. Η Ουκρανία διανύει μια πολύ δύσκολη περίοδο. Η Ουκρανία πραγματικά χρειάζεται ένα σταθερό εταίρο γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να καταγράψει κάποια πρόοδο. Η συνεργασία με την Eurojust είναι κάτι σημαντικό για την Ουκρανία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά το Μαυροβούνιο, σε Βούνιο, ως υποψήφια χώρα της Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύνευση αυτή τη συμφωνίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό βοηθάει την ενσωμάτωση της χώρας στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συμβάλλει στο να προετοιμαστεί η χώρα για την μελλοντική της ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σύντομος. Η Άννα παρακαλώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω εδώ. Θέλω παρακαλώ να σας ρωτήσω πώς τα καταφέρατε επιτυχώς να πείσετε συγκεκριμένες χώρες μέλη να συνεργαστούν όταν μιλάμε για επίπεδο ε, δικαστικής αρρωγής. Ε, εδώ ε, αντιμετωπίστε και το θέμα της διαφοράς. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, οι ίδιοι οι εισαγγελείς λένε ότι δεν κατάφεραν να επιτύχουν πλήρη συνεργασία ε, για περιπτώσεις ε, διαφοδοράς με τους Γερμανούς ε, για πωλήσει υποβρυχίων. Ενώ στην Γερμανία έχουν καταδικαστεί άτομα για δωροδοκία αξιωματούχων στη χώρα μου. Αυτή η συνεργασία υπάρχει γιατί έγιναν συμφωνίες στην Γερμανία μεταξύ των εισαγγελέων και των ε, Υπέτειο για, για ότι θα αποκαλύψουν ε, τους διεφθαρμένους στη χώρα μου και ενδεχομένως και στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια περίπτωση στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ. Γιατί μιλάμε λοιπόν. Γιατί μιλάει το Συμβούλιο σε αυτή την απόφαση όταν παράλληλα Αφήνουμε τις χώρες μέλη σε ξεκάθαρες περιπτώσεις διακρατικής διαφθοράς να μην συνεργαστούν, να μην καλούνται να συνεργαστούν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα δίκτυο πληρωμών που έγιναν με διάφορους τρόπους. Και εκεί τίθεται το θέμα της ε, ε, του ξεπλήματος και της τρομοκρατίας. Ε, για την Ουκρανία θα ήθελα να πω ότι πραγματικά ελπίζω αυτό να είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ε, ε, Ουκρανία στην καταπολέμηση της διαφθοράς γιατί η καταπολέμηση της διαφθοράς στην ε, Ουκρανία συνδέεται με την καταπολέμηση της διαφθοράς της χώρας μας. Ε, Μισελ, την προηγούμενη φορά που είτε ήταν ιδιαίτερα πιεσμένο το χρονοδιάγραμμά μας εδώ το πρώτο θέμα είναι η αντιτρομοκρατία Υπήρχαν ε, ερωτήσεις από την Επιτροπή, από τα μέλη και αυτό είναι κάτι που πιέζει. Μήπως θα μπορούσες να απαντήσεις πρώτα σε αυτές τις ερωτήσεις όσο γίνεται πιο σύντομα. Δίχως άλλο θα οργανώσουμε την επόμενη επίσκεψή του στην Επιτροπή και ελπίζω ότι τώρα θα είναι πιο χαλαρά τα πράγματα και θα έχεις περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σου. Θερμή παράκληση να είσαι σύντομη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση σας, κυρία Κάφμαν, και όντως ε, σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη, αυτό που αναφέρατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το NCS ε, είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ένα δίκτυο. Είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Να υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο να ξεπερνά τα υπόλοιπα δίκτυα της Τρομοκρατία. Το άρθρο 12 και 13 λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά και βλέπουμε σταδιακά ιδιαίτερα τα και 10 χρόνια στην τρομοκρατία. Το 2005 υπήρχε αυτή η υποχρέωση της ε, απόφαση του Συμβουλίου του 2005 που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να παρέχουν πληροφορίες στη Eurojust. προσκαλώντας ε, τακτικά τους υπευθύνους της Eurojust και με όλες τις δράσεις είδαμε λοιπόν ότι είμαστε στην κορυφή ε, των θεμάτων αυτών σε ό,τι αφορά την συνεργασία και τα στρατηγικά ζητήματα. Αυτό λοιπόν είχε να κάνει με την απόφαση του Συμβουλίου 2008 2018-2013. Τώρα λοιπόν προσπαθούμε τουλάχιστον μιας και έχει συσταθεί το ENCS, να επικεντρωθούμε σε αυτές τις τρεις προτεραιότητες. Αλλά φυσικά οι δικαστές σε πολλές χώρες έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας και αυτό είναι επιπλέον προς τα κοντά τους. Λοιπόν, πρέπει να διοργανώνουν και οργανώσεις και συναντήσεις και το καθεξής. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχουν ειδικέ συναντήσεις με τα άτομα αυτά για να δούμε του τι θα πρέπει να περιληφθεί από στρατηγική άποψη τις πραγματικές προτεραιότητες. Άρα χρησιμοποιούμε κάθε πρωτοβουλία και οποιοδήποτε βήμα μπορούμε να κάνουμε προκειμένου τα δίκτυα να είναι ανώτερα από τα υπόλοιπα δίκτυα. Και αυτό είναι ουσιαστικά ο λόγος ύπαρξης του ENCS. Ε, για την Ουκρανία, για το σχέδιο συμφωνίας, για το JSP, όντως ήταν θετικό για το ότι συμπεριλαμβάνονται τα θέματα προστασία των δεδομένων με την συμπεριληψή και ενός διαμεσολαβητή, ο οποίος φαίνεται ότι αποτελεί εχέγγυο για το Μαυροβούνιο. Καλό σημείο λοιπόν και αυτό. οι προτεραιότητε τώρα και το πώ διαμορφώνονται. Βάσει των εμπειριών μας, σε ποιες χώρες έχουμε μεγάλη εμπειρία. Στην Ουκρανία, προφανώς τα τελευταία 10 χρόνια, είχαμε 62 υποθέσεις για 25 συντονιστικέ συναντήσεις, κοινή ερευνητική ομάδα σε εξέχουσες υποθέσεις, υπήρχε για παράδειγμα για την ε, απάτη ΦΠΑ, το λαθρεμπόριο τσιγάρων, συνεργασία, τέτοια σημαντικά ζητήματα. Εφόσον υπάρχει συμφωνία δικαστικής συμφωνίας, συνεργασίας, όπως υπάρχει και με άλλες χώρες, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη δραστηριότητα και νομίζω ότι έτσι απαντάμε στο ερώτημα της κυρίας Γκρίσπεκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την ενθάρρυνση αυτή που μας ε, δίνετε, για τα λόγια αυτά που μας λέτε. Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει μία απάντηση για την ε, ποινική δικαιοσύνη, για την προσαγωγή των υπετίων και φυσικά τηρουμένων των προδιαγραφών του κράτους δικαίου. Δεν μπορώ λοιπόν παρά να συμφωνήσω με αυτά που μας είπατε. Σας είπα πώς διαμορφώνονται οι προτεραιότητες και αυτά λοιπόν μπορεί να τα εφαρμόσετε και για το Μαυροβούνιο για το οποίο είσαστε εισηγήτρια. Είναι τμήμα των Δυτικών Βαλκανίων και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχουν υπάρχει πραγματική ανάγκη να προσεγγίσουν τα Δυτικά Βαλκάνια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υποψήφιες χώρες και όντως σε σχέση με το Μαύρο Βούνιο δεν βλέπουμε να αποτυπώνεται αυτό στον αριθμό των υποθέσεων. Έχουμε μόνο 10 υποθέσεις που δεν ε, αναφέρθηκαν στις συναντήσεις συντονισμού, αλλά όπως έχει η κατάσταση σήμερα με την ασφάλεια, πραγματικά θα πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για το Μαυροβούνιο και σε ό,τι αφορά τους ραταπούς μαχητές κατά τον... Ε, εμπορίων των, της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και ούτω καθεξής. Και αυτό θα έχει ύψιστη σημασία. Με τη Ρωσία γίνονται διαπραγματεύσεις. Δεν έχουν ε, ακόμα περατωθεί για λόγους ε, προστασίας δεδομένων. Βεβαίως ε, έχουμε κάθε διάθεση σε καθεστώς απόλυτης ε, διαφάνειας να μοιραστούμε με εσά τα στοιχεία που έχουμε για το αφορά την τρομοκρατία και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Υπάρχει η 7η Συμφωνία Συνεργασίας. Υπάρχει συνεργασία της Νορβηγίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελβετίας τα αποτελέσματα της ε, συνεργασίας είναι πάρα πολύ καλά και πραγματικά αυτό επηρεάζει και τον αριθμό των περιπτώσεων και την ποιότητα των περιπτώσεων. Να σας ε, δώσω ένα παράδειγμα. Συντονίσαμε μία περίπτωση το 2013 χάρη στη βοήθεια των δικαστών της Νορβηγίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και πραγματικά ε, υπήρξε μεγάλη προστιθέμενη αξία. Είχαμε και ένα κέντρο συντονισμού Στις 12 Νοεμβρίου έγιναν πολλές συλλήψεις και αυτό έγινε σε στενή συνεργασία με την Ελβετία και την Νορβηγία. Όπως σας είπα, είναι θέμα και αριθμού και ποιότητας περιπτώσεων. Um, uh, in... Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της Ουκρανίας και του Μαυροβουνίου. Αναφέρθηκαν ορισμένες περιπτώσεις απάτης, ξεπλήματος, ε, διαφθοράς στην Ουκρανία. Πράγματι υπάρχει ανάγκη για δικαστική συνεργασία. Τώρα Α, επανέρχομαι στο τελευταίο ερώτημα της κυρίας Άννας Γκόμες. Εμείς θα πρέπει να πείσουμε τις χώρες μέρη να κάνουν καλύτερη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από την Eurojust. Εμείς παρέχουμε μία υπηρεσία, εργαζόμαστε με βάση το αίτημα που θα μας υποβληθεί Υπάρχει το άρθρο 85 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο αυτό παρέχει περισσότερες δυνατότητες ανάληψη πρωτοβουλειών. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να το ξανασκεφτούμε αυτό το θέμα γιατί όλες οι χώρες μέλη με ενθουσιασμό ζητάνε να τους δοθεί βοήθεια και αυτό σε ό,τι αφορά ορισμένε δοφέ εγκλήματο. Μπορούμε να του βοηθήσουμε, ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα, αλλά είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε γρήγορες λύσεις, να αντιδράσουμε άμεσα. Γι' αυτό το, το λόγο έχουμε δημιουργηθεί και γι' αυτό το λόγο πολεμάμε. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ε, καλός, ωραίος ο τρόπος που τελειώσατε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ως πρόεδρο τη Eurojust για την επίσκεψή σας. Ευχαριστώ και τους εισηγητές για την παρουσίασή τους. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που πήραν μέρος σε αυτή τη συνάντηση. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 16 Δεκεμβρίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα γιατί οι διερμηνείς θα πρέπει να φύγουν, έχουν συγκεκριμένο ωράριο. αν θα την τον στον Σεράιο. Σημείο 24α. Στις 9 Απριλίου ο κύριος Ράιασον ε, υπέβαλε ένα γραπτό ερώτημα στην Επιτροπή σχετικά με την μεταγραφή των μέτρων ε, προλυσαβών στην σε ό,τι αφορά τη συνεργασία ε, στην αστυνομία και στο δικαστικό κλάδο. Η απάντηση από την Επιτροπή στις 19 Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με τον κανόνα 130, ζητήθηκε το ερώτημα να συμπεριληφθεί στη ημερησία διάταξη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, η οποία συναντήθηκε για μια ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή. Επιτρέψτε μου να δώσω το λόγο του κυρία Κοράντο και μετά στα μέλη που θα επιθυμούσαν να πάρουν το λόγο. Η Άννα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπουμε τελευταία ότι παρατηρείται μία αύξηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού καθώς και των εγκλημάτων που οφείλονται σε αυτό. Αυτό είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Αυτό είναι κάτι που είδαμε τώρα τελευταία. Αυτό είναι κάτι που απειλεί τη δημοκρατική μας κοινωνία. Η απόφαση της Επιτροπής είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που απαιτούνται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση. Διάβασα την έκθεση Επιτροπής και καθίσταται σαφές ότι υπάρχουν κενά στις διάφορες χώρες. Παρατήρησα ότι αυτό ισχύει σε ό,τι αφορά τάσεις ξενοφοβίας και ρατσισμού καθώς και για τα εγκλήματα που γίνονται στο όνομα, στο όνομα αυτών. Θα πρέπει να υπάρξουν διμερείς διαλογοί μεταξύ των χωρών μελών. Δίχως άλλο υπάρχουν πάρα πολλά κενά θα πρέπει να προωθηθεί η ιδέα του διμερούς ε, διαλόγου. Η Επιτροπή θα έπρεπε να μας πει σε τι σημείο βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της απόφασης ε, πλαίσιο. Εάν το θέμα αυτό δεν έχει επιληθεί, δεν είστε ενδεχομένω η στιγμή για να ξεκινήσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα μίσους κατά της κοινότητας στο ΛΟΑΔΑ. Τα μέλη της κοινότητας στο ΛΟΑΔΑ ε, ε, είναι όλο και συχνότερα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων. Το θέμα είναι αν θα μπορούσε η Επιτροπή να, δει, την τη δυνατότητα να επεκταθεί η απόφαση πλαίσιο και σε φυσικές περιπτώσεις. Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, ε, αναφορά σε μία αναθεώρηση. Πότε θα γίνει μία αναθεώρηση της οδηγίας, ενδεχομένω από μέρου της Επιτροπής, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρχει και ε, μία ε, νομοθεσία σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Σας παρακαλώ να αναφερθείτε άμεσα στο θέμα αυτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους, ε, ε, την ευκαιρία που μας δίνετε να απαντήσουμε τις, ε, στην προφορική ερώτηση και όπως είπατε, όντως αυτό υπογραμμίζει, έχει υπογραμμιστεί αυτό το θέμα μάλλον αυτό και δεδομένη της μεταναστευτικής κρίσης και των τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη, η ξενοφοβία και ο ρατσισμός και πώς αντιμετωπίζονται δεδομένης και της ε, ε, εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Αυτό λοιπόν αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για την σωστή εφαρμογή του εργαλείου αυτού και έχει δηλώσει σε διάφορες περιστάσεις ότι δεν θα αντιστάσει να χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητες που της προσδίδει η συνθήκη μετά την ε, η υιοθέτηση της έκθεσης του 2014 για την εφαρμογή του ε, μέσου αυτού που αναφέρεται και στην προφορική ερώτηση και με σκοπό την προσαρμογή μετά τη μεταβατική περίοδο της Συνθήκης της Λισαβόνας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ανταλλαγή απόψεων με τα κράτη-μέλη εκφράζοντας ε, τις ανησυχίες της για την εφαρμογή της απόφασης πλαίσιο και για να ζητήσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις από τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει σημειώσει θετική πρόοδο σε διάφορες χώρες σε ό,τι αφορά και την προσαρμογή του ποινικού δικαίου προκειμένου να συνάδει με την απόφαση πλαίσιο εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία ανησυχίας και λαμβάνοντα υπόψη και τις διμερείς ε, επαφές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εφαρμόσει διαδικασίες ε, τις διαδικασίες που προηγούνται τις διαδικασίες στην παραβάση. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των συγκεκριμένων κανόνων επιτόπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αναφέρεται και στα συμπεράσματα του πρώτου εγγράφου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα συστήσει μια ομάδα για την ξενοφοβία που, όπου θα συναντηθούν οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και τη κοινωνία των πολιτών για να ανταλλάξουν ε, βέλτιστες πρακτικέ και να φροντίσουν ότι θα υπάρξει σωστή εφαρμογή και τη Ευρωπαϊκή και τη Εθνική Νομοθεσία στον τομέα αυτό. Σε ό,τι αφορά την ε, καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους και ε, εγκλημάτων που έχουν να κάνουν με το φύλλο και τον σε προσανατολισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό δεν είναι εφικτό δεδομένου του πρωτογενού δικαίου του, της Ένωσης. Ωστόσο, όλες οι δραστηριότητες που εκτελεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρέχει άρρωγη προς τα κράτη-μέλη έχουν να κάνουν και με την καταπολέμηση των εγκλημάτων και των ομιλιών μίσους. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και τη διάσταση του, του φύλου γιατί καλύπτονται ήδη από την νομοθεσία για τα εγκλήματα, για τα εγκλήματα μίσους και τις ομιλίες μίσους και σε ό,τι αφορά άλλους τύπους ε, εγκλημάτων. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Ο σκοπός της ερώτησης αυτής είναι να βρούμε γιατί δεν απαντήσατε όχι να επισέλθετε σε επίπεδο λεπτομέρειε τέτοιο και δεν έχουμε και χρόνο γιατί έχουμε και άλλο ένα θέμα. Σα παρακαλώ, περιτρέψτε λοιπόν στο θέμα αυτό, γιατί δεν απαντήσατε. Και θα ήθελα να διαβιβάσετε στην Επιτροπή. Έγραψα και στον Αντιπρόεδρο ε, Τίμερμαν, στον Επιτροπό Γιούροβα και Αβραμόπουλα, ότι θα πρέπει οι ερωτήσει να απαντώνται εγκαίρως, γιατί έχουμε 15 συζητήσει οι οποίε εκκρεμούν για ακριβώ λόγω των καθυστερήσεων αυτών. Τι για το θέμα λοιπόν αυτό και θα θέσω λοιπόν το θέμα αυτό και στην επόμενη προφορική ερώτηση. Αλλά σας παρακαλώ σε αυτή την ερώτηση να μα απαντήσετε γιατί δεν απαντήσετε εντός του χρονικού ορίου των 6 εβδομάδων. 15 συζητήσεις αναστήλαμε λόγω της καθυστέρησης. Καταλαβαίνουμε τι έχει το θέμα αυτό. Γι' αυτό θέσαμε το θέμα. Δεν χρειαζόμαστε περιγραφή. Το σημαντικό είναι γιατί καθυστερήσατε. Η κυρία Χέντε θεωρεί ότι απαντήθηκε στο ερώτημα του γιατί δεν ε, απάντησε η Επιτροπή μέσα σε 6 εβδομάδες. Ένα ναι ή ένα όχι. Όχι. Όχι, δεν μας δόθηκε κάποια απάντηση στο ερώτημά μας. Δηλαδή τα γιατί δεν, ε, δεν απαντήθηκαν. Όχι, όχι, δεν μας ικανοποιεί η απάντηση. Ωραία, θα περάσουμε στο επόμενο σημείο Κύριε Κοράου. Οι θα πρέπει να σταματήσουν στις 12.30. Κοιτάξτε, ε, θα ήθελα να απευθυνθώ στην Επιτροπή ότι δεν μπορεί να διεξαχθούν περαιτέρω συζητήσει. Το θέμα θα έπρεπε να απαντηθεί μέσα σε έξι εβδομάδες. Περνάω τώρα στο ερώτημα του κυρίου Κοράου που αφορά την μεταγραφή των μέτρων προ Λισαβόνας το αίτημα από την Επιτροπή στις 19 Νοεμβρίου 2015, εκτός δηλαδή της προθεσμία των 6 εβδομάδων, όπως καθορίζει ο κανόνα 130. Ο κύριος Κοράο, παρακαλώ. Το όσο γίνεται πιο σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήδη το Φεβρουάριο του 2015 υπέβαλα ένα ερώτημα με την υπογραφή και άλλων βουλευτών και ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει πότε θα είχε ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τη σωστή μεταγραφή των μέτρων δικαστική και αστυνομική συνεργασία όπω ενεκρίθηκε τη Συμφωνία Λισαμόνη. Τα μέτρα αυτά είναι δεσμευτικά από το 2014. Η Επιτροπή απάντησε ότι είχε δώσει προθεσμία στι χώρε μέλη για να εφαρμοστούν τα μέτρα μεταγραφή. 15η Μαΐου 2015 μετά την κοινοποίηση η Επιτροπή θα έπρεπε να προβεί στις αξιολογήσεις ετώντας από τις χώρες μέλη ε, να ε, συμμορφωθούν και ενημερώσει το Κοινοβούλιο. Στο τέλος Αυγούστου ε, επικοινώνησα με την Επιτροπή για να δω τι είχε γίνει από πλευρά τη. Τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συνομοθέτης θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Η απάντηση της Επιτροπής ε, ε, έφτασε καθυστερημένα και είναι εντελώς ανεπαρκής. Ε, δεν υπάρχει κατάλογος των μελών που έχουν καθυστερήσει, που δεν συμμορφώθηκαν. Δεν γνωρίζουμε την ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσουν, θα ληφθούν μέτρα κατά των χωρών μελών. Δεν γνωρίζουμε πότε η Επιτροπή θα ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά λοιπόν είναι αρμοδιότητε τη Επιτροπή, η οποία ενημερώθηκε από το 2009 ότι από την 1η Δεκεμβρίου του 2014 θα έπρεπε να ασχοληθεί με την εποπτεία. Το θέμα αυτό πολύ συχνά αντιμετωπίζεται ως θέμα δευτερεύουσα σημασία. Σήμερα όμως είναι στο καθημερινό χρονοδιάγραμμα της Ένωσης ω μέλο τη Επιτροπή Λίμπελ θα πρέπει να πετήσω κι εγώ κι εσείς κύριε Πρόεδρε μια συγκεκριμένη απάντηση. Δεν μπορούμε να μην έχουμε συγκεκριμένες αναφορές. Αυτό ακριβώς θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι αναμένουμε από την Επιτροπή. Θα ήθελα παρακαλέσω ο από της Επιτροπής να απαντήσει στα όσα ανέφερε ο κύριος Κοράου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη που μας δίνετε δυνατότητα να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Και ζητούμε συγγνώμη και για την καθυστέρηση στην υποβολή γραπτής απάντησης. Πράγματι, στο κεκτημένο του πρώην τρίτου πυλώνα συμπεριλαμβάνει πολύ, ένα πολύ σημαντικό φάσμα ε, νομικών μέσων στους τομείς ε, αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας. Και η κατάλληλη ε, και σωστή εφαρμογή του είναι θεμελιώδης σημασία ε, για την ε, προάσπιση των κρατικών ελευθεριών. Τα όσα υιοθετήθηκαν στις 28 Απριλίου 2015 υπογραμμίζουν ακριβώ αυτό. Όλες οι πράξεις που είναι νομικά ισχύουσε και δεσμευτικέ πρέπει να εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή έχει διασφαλίσει ότι μόνο τα έντεγα μέσα τα οποία είναι ενισχύ θα πρέπει να υλοποιούνται. Το δεύτερο εξάμεινο του 2014 κάναμε μια, ένα εγχείρημα χαρτογράφηση όλων των μέσων υπό τον τέταρτο πυλώνα και έτσι έχουμε εντοπίσει ε, νομικά μέσα που έχουν ε, εξαντλήσει τις νομικές προεκτάσεις και καλέσαμε την κατάργησή τους και η ΛΥΜΠΕ ενέκρινε ε, την έκθεση την περασμένη εβδομάδα και αυτό ανοίγει και το δρόμο για, το, για τα υπόλοιπα μέσα. Ασκήσαμε και το νόμο καθήκον παρακολούθηση της υλοποίησης ε, του κεκτημένου του πρώην τρίτου πυλώνα και ζητήσαμε από τα κάτι μέλη επισήμως να κοινοποιούν μέτρα εθνικής εφαρμογής. Ε, έχουμε μεταφέρει μια σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου. Αρχικά η προθεσμία ήταν 15 Μαρτίου, αλλά κατόπιν συζητήσεων με τα κράτη-μέλη έχει επεκταθεί έω τι 15 Μαΐου. Η προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ε, να ολοκληρώσει το κατάλογο κοινοποιήσεων, συνδράμοντα έτσι τα κράτη-μέλη όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Σε αυτό το στάδιο τη διαδικασία μπορούμε να πούμε ότι ορισμένα μέσα δεν έχουν μεταφερθεί πλήρω. Όμω, τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να στέλνουν κοινοποιήσει ε, των ε, μέτρων ε, μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Για την Επιτροπή, η πλήρη εφαρμογή από τα κρατημέλη είναι απαραίτητη για να ολοκληρωθεί η Ευρωπαϊ... ο ευρωπαϊκό κοινό χώρο δικαιοσύνη και να είναι ένα εύρωστο χώρο ενάντια στι απειλέ. Όλα αυτά θα βοηθήσουν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί καταλήλω ε, την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε αυτόν τον τομέα. Αυτό είναι ιδιαίτερα επίκαιρο δεδομένων και των ε, επιθέσεων στο Παρίσι και η Κομισιόν πράγματι ενισχύει τι προσπάθειέ τη ε, για να παρακολουθεί στενά την υλοποίηση. Η συνεργασία και τα αλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να βελτιωθούν. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναφέρει ότι μπορεί να αξιοποιήσει την αρμοδιότητα που δίνεται υπό τη συνθήκη ε, να εξετάσει ζητήματα μη κοινοποίηση και μη συμμόρφωση και να κινήσει και διαδικασίε υπεραβάσεω από αυτόν απαραίτητο. Η Κομισιόν θα εξακολουθήσει να παράσχει πληροφορίε ε, προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μέσω των υφιστάμενων διόδων και σημειώνουμε και το αίτημα να δίνουμε περισσότερε λεπτομέρειε όπου αυτό είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ. Κύριε Κορά, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να σχολιάσουν. Πιστεύω ότι η απάντηση συνεχίζει να είναι γενική. Είναι νεφελώδης και οι μεροφινίες και οι κατάλογοι. Η Επιτροπή για μία ακόμα φορά μας λέει ναι ασχολούμεθα, ναι με ποιους, με ποιες χώρες, ε, τι ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πολύ γενικά όλα αυτά. Για το Κοινοβούλιο δεν είναι αποδεκτές αυτές οι γενικότητες. Δεν με ικανοποιεί καθόλου η απάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αγιαλόπε. Πολύ σύντομα ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο και δεν έχει νόημα να επιμένουμε, αλλά δεν θα ήθελα να περάσει απαρατήρητο, γιατί είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας τεράστιος φορέας, ε, γραφειοκράτες, τεχνοκράτες, υπάλληλοι, σύμβουλοι, αλλά πάνω απ' όλα είναι πολιτικό θεσμικό όργανο, το οποίο είναι υπόλογο απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και έχει έρθει η ώρα όλα αυτά να τα παρατηρήσουμε, να τα προσέξουμε. Αυτές τις συνήθεις πρακτικές, ε, να μην απαντούν, να δίνουν κάτι γενικό απαντήσεις και τίποτα παραπάνω, χωρίς ε, συναφή στοιχεία, όταν μιλούμε για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που θα πρέπει να ασκήσει το κοινοβούλιο, πρέπει να σταματήσουν λοιπόν αυτές οι πρακτικές και να μην μάθαμε τα λόγια μας αυτό το ζήτημα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και τους δύο συναδέλφους. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε, και αυτό δεν ε, το απευθύνουμε σας προσωπικά, είστε εκπρόσωπος της Κομισιόν, είναι ότι διαμορφώνεται ένα πρότυπο όπου πρέπει να έχουμε χρόνο εμεί για να θεωρήσουμε αυτά τα στοιχεία. Ε, το θέμα δεν είναι αν θα δίνετε γενικόλογες απάντηση ή όχι, αυτό είναι δικαίωμά σα. Όμως, πρέπει να τηρείτε το χρονοδιάγραμμα. Γιατί αλλιώς μας αναγκάζεστε να θέτουμε ζητήματα στην μέσα διάταξη, ενώ δεν έχουμε τον χρόνο. Δεύτερον, οι εκπρόσωποι της Κομισιόν έρχονται εδώ και προσπαθούν να απαντήσουν πολύ γενικόλογα τις ε, ερωτήσεις που θα έπρεπε να είχαν πάρει τον χρόνο να τις απαντήσουν διεξοδικά. Και όπως λέει και ο κ. Λόπας έχετε τους πόρους για να απαντήσετε σε κάποια στοιχεία. Αυτό που ανέφερε η Άννα παράδειγμα. Ότι υπάρχει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχετε και τον χρόνο να το πράξετε. Και τέλο περιμένουμε γραπτή απάντηση από τον Αντιπρόεδρο και του δύο επιτρόπους ε, στην επιστολή μου, όπου τους ε, ρώτησα γιατί δεν γίνονται σε αυτά όλα αυτά και γιατί ω εκ τούτου πρέπει και εμεί να διοργανώνουμε τόσε πολλέ συζητήσει. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο που θα πρέπει και εσεί να το αντιμετωπίσετε, γιατί δεν γίνεται να συνεχίσουμε να έχουμε τις συζητήσεις αυτές στην εμείς διάταξη, να κάνουν οι προβουλευτέ τις ερωτήσεις και να συνεχίζετε αυτή η διαδικασία επάπειρων. Αν μπορείτε να διαβεβάσετε αυτές τις παρατηρήσεις θα ήμουν ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Sorry, any other business. Ναι, διάφορα. Εντάξει, τέλος συνεδρίαση.